to have you here. because we're getting off. Okay. Welcome back to... Ξεκινούμε τις εργασίε μας σήμερα το απόγευμα με το σημείο 10. Ε, με τα σημεία 10, 11 και 12. Κοινή συζήτηση. Το πακέτο κυβέρνου ασφάλειας την έκθεση για την φύση των απειλών, απάντηση στο εξελισσόμενο περιβάλλον των απειλών από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορική, την ΕΝΗΣΑ όπω την ξέρουμε όλοι. Μετά έχουμε το σημείο 11, το, το Κέντρο για τα Εγκλήματα στον χώρο τη Europol και το σημείο 12, δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στον χώρο. Θα ακούσουμε την παρουσίαση του προσκεκλημένου μας κύριου Steve Purser, επικεφαλής της τεχνικής υπηρεσίας της ΕΝΙΣΑ, τον Charles Έρτινγκ, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο και την παρουσίαση από τον κύριο Πολ Τίμερ, Διευθυντή Βιώσιμης και Ασφαλούς Κοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης ΚΝΕΚΤ της Επιτροπής. Στις 7 Φεβρουαρίου η Επιτροπή υιοθέτησε αυτό το πακέτο κυβέρνου ασφάλεια. Είχαμε μια ενημέρωση και από τους επιτρόπους ε, κύρια Κρούς και κύρια Μάρστρομ. Ένα σημαντικό έγγραφο που είναι σημαντικό για τις εργασίες της ΛΥΜΠΕ, την εσωτερική ασφάλεια, τον κυβέρνο έγκλημα, την προστασία των δεδομένων. Θα έχουμε μια κοινή συζήτηση μετά την παρουσίαση και από την ΕΝΙΣΑ και από την Europol και λίγο χώρο για συζήτηση. Είναι εδώ οι προσκεκλημένοι μας, τους καλωσορίζω τον κύριο Πέρσε, τον κύριο Έρτινγκ, τον ακούσαμε και το πρωί και τον κύριο Τίμερς. προτείνω να ακούσουμε τις παρουσιάσεις τους. Έχουμε μια μισή ώρα. Θα μπορούσαν να μιλάνε δεκάλεπτα ο καθένας και μετά να ξεκινήσει η συζήτηση. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Πέρσερ από την Ενίσα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που με καλέσατε εμένα και την ενίσχυα δηλαδή στο πρόσωπό μου. Θα σας μιλήσω για την ε, μελέτη της ενίσχυας, για την εξέλιξη των απλών. Εισαγωγικά. Η ενίσχυα είναι συνεργασία, όπως ξέρετε. Το business model μας στηρίζεται στη συνεργασία με άλλους, σε επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της Ένωσης ή και με τον ιδιωτικό τομέα. Ό,τι κάνουμε, γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, δεν είναι δική μας, αλλά κοινή δουλειά. Και αυτό που παρουσιάζουμε είναι το αποτέλεσμα του διαλόγου με τις διάφορες πλευρές. Τα περισσότερα από τα αποτελέσματα προέρχονται από τις βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες που υπάρχουν σε διάφορα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό διότι αυτό είναι ο τρόπο δουλειά μα στο μέλλον και στο κέντρο τη ε, συνεργασία μα με την Επιτροπή, όπου βλέπετε όλο ένα και περισσότερες διαστάσεις όπως ε, ΣΒΙΤ και εσωτερικέ επικοινωνίες. Δεν είναι λοιπόν δουλειά της ΕΝΗΣΑ αλλά όλων. Ξεκινώντας να σας πω ότι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε την επόμενη δεκαετία δεν είναι να λειτουργήσει διασυνοριακά η ασφάλεια σωστά, αλλά και, διακοινωτι... και Δηλαδή παρέχοντας ελευθερία ροή των πληροφορών μεταξύ των διαφόρων δομών για να μην γίνεται επικάλυψη δραστηριότητα και να μαθαίνουμε από τα λάθη ο ένας του άλλου. Και από την εμπειρία προφανώ. Ο κ. Στίμεν, ο κ. Ή ο εκπρόσωπος της Europol, τα συζητάμε αυτά σε τακτική βάση. Βεβαίως αυτό το μήνα βγάλαμε και τη στρατηγική, εκδώσαμε και τη στρατηγική για την ε, ασφάλεια της Ένωσης. Είναι ένα σημαντικό θέμα για την Ενίσσα που πιστεύω ότι θα μα βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα που θα προσπαθήσω να σα εξηγήσω εντάχει σήμερα. Το καλωσορίζουμε, θεωρούμε ότι είναι ένα μεγάλο βήμα μπρο. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν ξεκινήσω να σα λέω αυτά που θα σα πω. Ελπίζω να μην απογοητευτείτε, διότι είναι υψηλού επίπεδου παρουσίαση. Εγώ είμαι 18 χρόνια στην εμπροστοφυλακή των ε, δραστηριοτήτων και έχω πολλά και δεν ξέρω πολύ την τεχνική κατάσταση, κάτι το οποίο μπορεί να σας δυσκολέψει γιατί πρέπει να ξέρεις τα τεχνικά θέματα. Να προσπαθήσω να αλλάξω τα slide μου, δεν ξέρω αν θα με βοηθήσετε. we go. There we go. Thank you. So I'm going to give very brief... Να σας κάνω μια εισαγωγική παρατήρηση για την ενίσα. Κάποια εισαγωγικά σχόλια, την αρχική έκθεση και το, για το περιβάλλον απειλών, το βασικό θέμα, τα κύρια ευρήματα και κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, είμαστε νέα υπηρεσία σχετικά, το 4 δημιουργηθήκαμε. Έχουμε ένα, μας λένε κέντρο εμπειρογνωμοσύνης, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν το εννοούμε με την έννοια των σοφών, αλλά βασικά αντλούμε την εμπειρία από αλλού Χρειάζεται ωστόσο και κάποια εμπειρία για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο ρόλος μα είναι όχι μόνο να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή, αλλά να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ένα μεγάλο τμήμα τη δουλειά μα και ένα μεγάλο τμήμα των αποτελεσμάτων που θα δείτε σήμερα προέρχονται προφανώ από την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα. Εισαγωγικά, θα σας δείξω κάποιες εικόνες του πώς φαίνεται το περιβάλλον απειλών από την οπτική άποψη της ΕΝΗΣΑ. Λάβετε υπόψη βέβαια ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται οι απειλές είναι σύνθετος τρόπος, εξελίσσονται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Ένας για παράδειγμα είναι το πόσο αποφασιστικότητα έχουν οι αντίπαλοι σου, τι τους κινητοποιεί, τι ιδέες έχουν. Δεν είναι εύκολο να μελετήσουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλές μεταβλητές και τα στοιχεία ακόμα να έχουμε είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντομίσουμε τέτοιες απειλές. Τα τελευταία 20 χρόνια δουλεύω στον τομέα αυτό όπως σας είπα. Ο κλάδος θεωρεί ότι δεν υπάρχει μεγάλη σταθερότητα. Ένα παράδειγμα. Ξέρετε το Stuxnet, ξέρετε ότι αυτό άλλαξε, δεν άλλαξε σημαντικά, αλλά αυτό που άλλαξε ήταν ο στόχος αντί να μιλάμε για οικονομικές ζημιές, μιλάμε για ζημιές, για απώλειες ανθρώπους στον ανθρώπινο παράγοντα. Όπως το μετρολογικό δελτίο είναι. Όσο πιο μακριά είναι ο χρόνος, τόσο πιο αβέβαιη είναι η πρόβλεψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ε, ε, τις πληροφορίες που έχουμε, όπως ακριβώς και για τις περιπτώσεις μετεωρολογικού βελτίου. Τώρα, η ικανότητα αντίδρασής μας στον τομέα είναι καλός και μπορούμε να αποφύγουμε μεγάλες επιθέσεις. Δεν θα πρέπει να σας δημιουργούνται ανησυχίε εδώ, αλλά λάβετε υπόψη ότι οι δυνατότητες πρόβλεψης που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλές και θα παραμείνουν χαμηλές. Πρέπει να μπορέσουμε να αντέξουμε και να ζήσουμε με αυτούς τους περιορισμούς. Έχουμε και οι οικονομικές ε, πιέσεις έχουν, ε, οι επιτιθέμενοι διαπιστώνουν ότι έχουν καταλάβει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αδύνατα σημεία διότι εμείς δεν έχουμε δυνατότητα αντιμετώπιση σε ταχύτερο τρόπο και με μεγαλύτερη οικονομική δύναμη τις απειλές του Στην πραγματικότητα, καθώς ε, απαιτεί η επιχείρηση μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, είναι όλο και πιο δύσκολο να υπάρξουν σωστοί έλεγχοι. Αυτό το βλέπουμε παντού. Πρόκειται για μια ισορροπία που θα πρέπει να αντέξουμε. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστέ σε παγκόσμιο επίπεδο και άρα να εξισορροπήσουμε. Και αυτό δεν είναι το πιο ασφαλέ ή επισφαλέ, αλλά το, την ισορροπία μεταξύ των δύο. Η λύση βρίσκεται στην, στο συνδυασμό ανθρώπων, διεργασιών και τεχνολογιών. Α πούμε στην έκθεση. Η έκθεση αυτή καθεαυτή παρέχει μια εικόνα των απειλών και των υφιστάμενων και αναλυσόμενων και εξελισσόμενων τάσεων. Σημαντικό να τονίσω ότι τούτο δεν το κάνουμε εμείς. Δεν είναι δική μας η ανάλυση κινδύνου, απλά ε, συμπιλούμε μια σειρά αναλύσεων από άλλους. Και αυτό οικονομική διάσταση έχει. Εγώ με 30 ανθρώπους τι να πρώτο κάνω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε μια τέτοια δουλειά μόνοι μας, αλλά να ερμηνεύσουμε τη δουλειά που κάνουν άλλοι και να την περάσουμε στι κοινότητε με τι οποίε συνεργαζόμαστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν κάναμε ανάλυση περί των 100 εκθέσεων, πρόσφατων εκθέσεων από σειρά πηγών. Ποιο είναι, ποιος είναι ο, η ομάδα στόχο. Άνθρωποι που λαμβάνουν αποφάσει, ε, επαγγελματίε τη ασφάλεια, επαγγελματίε τη διαχείριση κινδύνων, άτομα σε υψηλό επίπεδο. Ε, η έκθεση μάλλον είναι υψηλό επίπεδο για να υπάρχει κατανόηση. Ε, Ξέρετε ότι έχουμε το μότο «Αν ξέρεις τον εαυτό σου, ξέρεις τον εχθρό σου». Οι χίλιες μάχες είναι χίλιες φορές γνώση. Δεν μπορούμε βέβαια να προβλέψουμε 100%. Είναι σημαντικό όσο να μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα και εκτίμηση του τι συμβαίνει για να, έχουν, για σας επιτρέπουν να λάβετε τις σωστές αποφάσεις. Μέθοδος. Συλλέγουμε και συνολοποιούμε τις πληροφορίες, τις συμπληρούμε σε μία ενιαία έκθεση. Όπως σας είπα, 120 εκθέσεις λάβαμε υπόψη, περισσότερες του 12. Σύγχρονη, επίκαιρη η πληροφόρηση λοιπόν. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν υφιστάμενο τοπίο απειλών, αναδιόμενο τοπίο απειλών. Τι είναι αυτό που μπορεί να ξεκινήσει να γίνει ή πρέπει να προσέχουμε αν είστε εσείς πρέπει να προσέχετε δηλαδή ως υπεύθυνοι λήψη αποφάσεων. Sorry. I'll go down a click for you. There we go. That's just a diagrammatic. Αυτό βλέπ, εδώ είναι μια υπομορφή διαγράμματος παρουσίαση που δείχνει τον τρόπο που δουλεύει το, η ενίσα στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να έχουμε ακόμα περισσότερες επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους καθιστώντας πιο αποτελεσματική τη διαδικασία. Δεν θα αναλύσουμε εμείς τους κινδύνους, θα αναλύουμε ίσως κενά, πιθανά κενά που εμφανίζονται στις εκθέσεις άλλων, αλλά στην, εν γέννη θα προσπαθούμε να να καθιστούμε όσο χρησιμότερο γίνεται την υφιστάμενη ενημέρωση για όλες τις κοινότητες λαμβανόντων τις αποφάσεις. Τα, τα κύρια ευρήματα. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, εντοπιστήκαν οι βασικές κυβερνόπηλες αυτή τη στιγμή με βάση τη συχνότητα. Όπως θα σας πω στο τέλος, ο αντίκτυπος είναι λίγο πιο δυσδιάκριτος και θα σας εξηγήσω γιατί. Οι τάσεις ε, προέρχονται, από τη σύγκριση της υφιστάμενης ε, ενημέρωσης για τις επιλές με αυτές των τελευταίων ετών. Και τέλος ε, διατυπώνουμε μια σειρά πιθανών αναδυόμενων απειλών. οι τομεί αυτοί ούτω ή άλλω υπάρχουν και στο πρόγραμμα τη Ένωση και στο δικό μα, οπότε δεν νομίζω ότι θα έχετε αντιρρήσει. Ε, κινητή, κινητές, κινητοί υπολογιστές, ε, κοινωνικές ε, τεχνολογίες κοινωνικών δικτύων, κριτικές υποδομές κλπ. Ποιες είναι οι κύριες απειλές συχνότητα. Πολύ γρήγορα θα σας τα πω, με πολύ ε, γενικευμένη πληροφόρηση. Ε, εκμετάλλευση της χρήσης των ιστοσελίδων στις οποίες μπαίνει, το drive-by exploit. Αν δεν, είσαι, αν δεν σωστά και μπει σε ένα site, μπορεί να σου αλλάξει το σύστημα και να κάνει τις στα μάτια στο κομπιούτερ σου. Είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε χρόνια. Η e, πολύ συχνή. Έχουμε προχωρήσει σε μια πολύ εξελιγμένη προστασία εις ε, χρησιμοποίηση κωδικών. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το SQL που έχει αδυναμίες για να ε, ενέσεις ε, οδηγίες στο κομπιούτερ που δεν υπάρχουν, εκμεταλλευόμενος δηλαδή το λειτουργικότητα του προγράμματος, κλέβοντας πληροφορίες και λοιπά κακά πράγματα. Ε, εργαλεία εκμετάλλευσης, botnet, τα ξέρετε, είναι μια σειρά, ένας τεράστιος αριθμός ε, διεφθαρμένων ε, ε, κομπιούτερ που χρησιμοποιούνται για να μπουν στο κομπιούτερ, άρνηση υπηρεσίες, φορτώνουν την, το μηχάνημα και όταν το φορτώνουν μπορείς να μπει μέσα. Το phishing που είναι τεχνική στον εκμετάλλευση των κοινωνικών δικείων. Πείθει τον κόσμο να σου δώσουν πληροφορίες για τους ίδιους που είναι εύκολο για να μπορέσεις μετά να μπει σε ένα σύστημα ή να κάνεις αγοραπολισίες στο ίντερνετ κατόπιν. Ε, χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών το logware και το scareware είναι ψεύτικα software ή ψεύτικες προειδοποιήσεις, θα σας μιλήσουν οι συνάδελφοι, έχουν καλά παραδείγματα. γίνεται και το spam. Κατάχρηση του email, το ξέρετε όλοι αυτό. Αυτή είναι η εικόνα. Ε, δεν νομίζω ότι μπορείτε να το διαβάσετε και ούτε καν θα προσπαθήσω να το αναλύσω γιατί στο δεκάλεπτο ήδη έχω αρχίσει και τελειώνει. Δείτε την έκθεση χωρίς να ξέρετε τεχνικά στοιχεία ή να έχετε εμπειρία. Αυτό που σας λέει το διάγραμμα με ωραίο τρόπο είναι πώς εξελίσσονται με το χρόνο οι απειλές αυτές. Γίνονται χειρότερες, γίνονται καλύτερες και πώς ε, περιγράφω και πώς χαρτογραφούνται στους διάφορους τομείς που προενέφερα. Μια εικόνα του χρόνου, ε, η εικόνα θα είναι διαφορετική, αλλά είναι καλό να ξέρουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Επίσης, προχωρούμε σε μία ανάλυση των ε, παραγόντων απειλής που, που σας λέει ποιοι είναι αυτοί που σας απειλούν και κάποιες φορές τα στοιχεία ε, είναι και εντυπωσιακά. Δεν ξέρω αν αυτά ταιριάζει με την εικόνα του πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η άλλη πλευρά δηλαδή του νομίσματος. Αυτοί που κάνουν τις επιθέσεις. Και μετά για κάθε τομέα που ανέφερα, αυτά είναι τα μεγάλα δεδομένα για παράδειγμα, δίνουμε λεπτομερέστερη ανάλυση των απειλών στο συγκεκριμένο τομέα. Η έκθεση είναι περί τις 100 σελίδες, μεγάλη έκθεση, αλλά μπορεί να διαβάσετε ό,τι σας αρέσει. Αν σας ενδιαφέρει το cloud ή τα κινητά, τόσο να διαβάζετε τα συγκεκριμένα τμήματα. Και, και έτσι μπορεί να μάθετε τι γίνεται στον τομέα αυτό. Συμπεράσματα. οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν απλά και φτηνά όπλα συνολικά. Δεν είναι αλήθεια πάντα. Το Stuxnet ήταν πολύ σοφιστή και κώδικας αλλά εν γέννη τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι εύκολα και εύχριστα και υπάρχουν για χρόνια. Επίση, για πολύ καιρό δεν διαπιστώνονται οι αδυναμίε του συστήματο. Παλιά, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, έρχομαι από ένα εμπορικό περιβάλλον με υψηλή προστασία και παρά τα αυτά τι τρύπε τι καλύπταμε μετά από μήνε, αρκετού μήνε. Υπάρχει ένα πρόβλημα τροτότητα δηλαδή, γιατί πρέπει να, εξισορροπεί την ανασφάλεια με τα κέρδη, τα πιθανά κέρδη του να σταματήσει τι επιθέσει, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε καλύτερα. Επίση, δεν ξέρουμε αρκετά για του επιτιθέμενου και τι τακτικέ που ακολουθούν. Η έκθεση δίνει κάποιε περισσότερε πληροφορίε γι' αυτό, αλλά δείχνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Και παρότι ότι γίνονται πολλά πράγματα στον τομέα τη συνεργασία, χρειάζεται πολύ, πάρα πολύ περισσότερη συνεργασία οι συστάσει. Να σα τα πω πολύ πιο γρήγορα από αυτά που τα λέω τώρα. Συλλέξτε και αναπτύξτε καλύτερα στοιχεία για τις, τους ε, τρόπους επιθέσεων ε, στη στρατηγική το είδαμε αυτό. Μεταξύ των άλλων ε, η, η, παραβίαση πιστοποιητικών ασφάλειας είναι πολύ χρήσιμη. Συλλέξτε και αναπτύξτε καλύτερα στοιχεία για τον αντίκτυπο που επιτυγχάνεται. Αυτό είναι δυσκολότερο. Όπω ξέρετε, οι επιχειρήσει δεν λένε ότι του έγινε hacking ή ότι τέλο πάντων επηρεάστηκε η επιχείρησή του με τον ΑΒ τρόπο, δεν είναι καλό. Και χρειάζεται, χρειάζεται να αναλύσουμε τον αντίκτυπο, γιατί αυτό δείχνει τη διαφορά μεταξύ μια σημαντική ε, δομή επίθεση και ενό και μια λιγότερη. Συλλέξτε και διατηρήστε περισσότερα ποιοτικά στοιχεία για του φορεί τη απειλή. Αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη. Παρά μόνο ίσω στην στρατιωτικό τομέα ή τι αντικατασκοπίε. Η ανάλυση των υπεύθυνων ε, επιθέσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένα, είναι σημαντικό κομμάτι στο puzzle και αλλάζει συνεχώ. Χρησιμοποιήστε κοινή ορολογία. Αυτό είναι σημαντικό όταν μοιράζεται κανεί πληροφορίε. Αν δεν χρησιμοποιείτε αντίστοιχου όμοιου όρου, και δεν χρειάζεται να είναι δρακόντιο, αλλά χρειάζεται να υπάρχει ένα επίπεδο συνεκτικότητα ε, για να μπορεί να εμπιστεύεται ο ένα τον άλλον και να ξέρει ότι οι πληροφορίε που δίνει είναι συγκρίσιμε διασυνοριακά και μέσα στην κοινότητα χρησιμοποιήστε την ε, προοπτική του χρήστη γιατί συχνά πολλή δουλειά γίνεται με βάση τους στρατιωτικούς ή ε, τους πανειδικού χρήστες και όχι τον, τον κανονικό χρήστη. Επίσης, ε, χρησιμοποιήστε ε, περιπτώσεις χρήσης των, του τοπίου Μαζέψτε, συλλέξτε επίσης πληροφορίες ασφάλειας. Αυτό είναι σημαντικό. Γίνεται, αλλά χρειάζεται περισσότερο. Πρέπει να ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, πώς, τι θα εμπλακεί και πώς θα αντιμετωπίσεις μια τέτοια εμπλοκή. Και όλος αυτός ο κλάδος χρειάζεται να ενωθεί για να έχει σωστά και κάντε αλλαγές στους ελέγχους ε, ασφάλειας. Πρέπει να πηγαίνουμε σε ελέγχους ασφάλειας ε, που θα προσανατολίζονται περισσότερο στα δεδομένα. Πριν από, πριν από 15 χρόνια έγιναν τα firewall. Ωραίο. Το τείχος ασφαλείας. αλλά τώρα, επειδή τον ανοίγουμε για να μπαίνουν οι υπεύθυνοι ασφάλειας της εταιρεία, ε, χρειαζόμαστε άλλους μηχανισμούς που θα ανταποκρίνονται στο πώς δουλεύουμε σήμερα. Αυτή ήταν η τελευταία ε, ε παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πούρσερ για την παρουσίαση μας κάνατε εξ ονόματος της ΕΝΙΣΑ όπου παρουσιάσετε το έργο του φορέα σας Πολλά χέρια σηκώθηκαν. Αλλά θα πρότεινα να, ακούσουμε, να ακούσουμε όλες τις παρουσιάσεις και μετά να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε αφού ακούσουμε και τον κύριο Ερτουρ, ο οποίος θα παρουσιάσει την άποψη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κυβερνεγκλήματος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ κάτω να λειτουργήσω τον υπολογιστή γιατί δεν δουλεύει από αλλού. <clears throat> σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα σας δώσω μια λιγότερο λεπτομεριακή και ίσως πιο γενική επισκόπηση του πώς βλέπουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Κύβερνο ανάπτυξη και εξέλιξη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο και περισσότερες χώρες θα καλωδιωθούν στην Ευρώπη είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, σε άλλες περιοχές όπως η Αφρική είναι μόνο 34% το επίπεδο αυτό. Βλέπουμε επίσης ότι το, ο κυβερνόχωρος θα ολοκληρώσει όλα τα δεδομένα μας και μετά θα δρά και εξ ονοματός μας. Αυτό δεν αφορά μονάχα τα δεν είναι τωρινό σε 10 χρόνια ή παραπάνω και μετά θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο διαδίκτυο χωρίς τον υπολογιστή μας και θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερους κινδύνους δυστυχώς. Το ίντερνετ θα γίνει δευτερεύον. <clears throat> Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά στο μέλλον θα γίνει δευτερεύον. Θα είναι απλώς ένας διευκολυντής επικοινωνίας και θα είναι σαν τον ηλεκτρισμό, ένα τμήμα του συνολικού πλαισίου. Θα είμαστε πάντα επιγραμμικοί, πάντα επιγραμμικοί. Γι' αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα όταν έχουμε νομοθετικέ πρωτοβουλίε, ότι αυτό δεν θα είναι κάτι το οποίο θα το επιλέγουμε. Θα είμαστε κολλημένοι στο διαδίκτυο πάντα. Πάντα τα ψυγεία μα, τα αυτοκίνητά μα, οι βηματοδότες μας, τα παιδιά μας, οι γάτες μας, όλοι αυτοί θα βρίσκονται στο διαδίκτυο συνέχεια. Περισσότερη καινοτομία λοιπόν ευμάρια, αν, ε, άνοδος, δημοκρατία, ελευθερία, γνώση, πιο απλή, πιο εύκολη ζωή, πιο ασφαλής ζωή, περισσότερη εκπαίδευση, αλλά θα αλλάξει και τον πόλεμο το μέλλον. Οι πόλεμοι μας ήταν πάντα πόλεμοι στην ξηρά, μετά ήταν στη θάλασσα, μετά ήταν στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, μετά στο διάστημα, αλλά μετά θα γίνει ο επόμενος πόλεμος στον κυβερνόχωρο. Και βλέπετε τις προετοιμασίες που γίνονται ήδη. Η κυβερνοκατασκοπία επίσης. Ο ψυχρός πόλεμος και η ανθρώπινη εμπλοκή στη συλλογή πληροφοριών θα αλλάξει ριζικά και θα δείτε να γίνεται ο κυβερνοπόλεμος και οι κυβερνοεκδιασμοί από το διαδίκτυο ο κυβερνοακτιβισμός επίσης και ο κυβερνοτρο... η κυβερνοτρομοκρατία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πατάει το κουμπί. Χρειάζονται περισσότερη, πολύ λιγότερη δύναμη και πολύ λιγότερη στρατιωτική δύναμη. Χρειάζεται μονάχα ένας υπολογιστής, καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο και να είναι κανείς πολύ καλός στα θέματα αυτά, καλός hacker. Αυτά δεν είναι τμήμα της εντολής του EC3. Τα αναφέρω γιατί σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυνατότητες μιας επίθεση προτού της αντιμετωπίσει. Θα πρέπει να καταλάβουμε <coughs> να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών συλλογή πληροφοριών, τη αστυνομία και του στρατού. Όταν πηγαίνω στο διαδίκτυο, μα ακολουθούν οι εγκληματίε. Υπάρχουν δύο μορφέ εγκλήματο. Το πραγματικό κυβερνό έγκλημα που μπορεί να γίνει μόνο στο κυβερνόχωρο και μετά το έγκλημα που διευκολύνεται από τον κυβερνόχωρο παραδείγματο χάρη οδηγεί σε εκμετάλλευση βιασμού παιδιών στον πραγματικό κόσμο, αλλά χρησιμοποιεί κανεί το διαδίκτυο για να μπορέσει να πουλήσει τι ταυτότητε αυτών των παιδιών επιγραμμικά. Τι βλέπουμε τώρα. Απάτες ΦΠΑ. Χάνει 160 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε απάτες ΦΠΑ. Τα 60 από αυτά, 60% από αυτά από το οργανωμένο έγκλημα και πάντα με ε, υπολογιστές. Οι, τα λίτρα τα οποία ζητούνται είναι μάλλον η σύλληψη, ναι, τα λίτρα τα οποία ζητάτε όταν κάποιος σας έχει μπλοκάρει τον υπολογιστή, έχει πάρει όλα τα δεδομένα σας και σας ζητάει να πληρώσετε. Μια μπίζνα 100 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία λειτουργεί πολύ καλά σε ορισμένα μέρη τη ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλές οι συμμορίες που κάνουν κάτι τέτοιο. Οι τρόε των τραπεζών είναι αυτοί οι οποίοι ε, ανοιχνεύουν τις ε, πληρωμές από το διαδίκτυο και υπάρχει επίσης και το σύννεφο, το νέφο. Ε, θα σας δώσει ο συνάδελφό μου μετά περισσότερες πληροφορίες, αλλά για, μένα θέλω να τονίσω δύο στοιχεία. Όλοι μας σύντομα θα έχουμε όλη την πληροφορία μας την προσωπική στο σύννεφο, στον νέφος Και θα πρέπει να ξεχάσουμε τα λάπτοπς και τους υπολογιστές γραφείου. Όλα τα δεδομένα μας θα είναι στο σύννεφο, στον νέφος και η αστυνομία θα έχει δυσκολία να βρει αυτές τις πληροφορίες γιατί οι εγκληματίες θα χρησιμοποιούν και αυτή τέτοια δίκτυα τα οποία θα μπορούν να υποκαθιστούν αυτό το δίκτυο θα αλλάξει τον έφος λοιπόν της ζωής μας. Επίσης θα αλλάξουν πολλά πράγματα γιατί αυτό το έγκλημα μπορεί να γίνει και από αλλού. Όταν βλέπετε παραγωγός την Αφρική να περάσει από το τωρινό επίπεδο στο 80% θα υπάρχει και περισσότερο έγκλημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τώρα η διαφορά μεταξύ του παραδοσιακού οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχουν γεωγραφικέ συνδέσει μεταξύ του εγκλήματο και του εγκληματία στον επιγραμμικό κυβερνό εγκληματικό χώρο. Είναι εύκολο για του ε, εγκληματίε να κάνουν εγκληματικέ ενέργειε χωρί να είναι παρόντες επιτόπου. Μπορείτε να είστε σε μια χώρα και να εγκληματείτε σε άλλε δέκα χώρε και κανεί δεν ξέρει τι κάνετε. Γιατί μπορείτε πολύ εύκολα να κρυφτείτε με πολλές υπηρεσίες που είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Είναι πολύ λιγότεροι πόροι που χρειάζεστε για να εγκληματίσετε και η αλυσίδα αξίας στον κυβερνόχωρο είναι πολύ πιο μικρή. Αν θέλετε να πουλήσετε κοκαίνη πρέπει καταρχήν να καλλιεργήσετε στην Κολομβία, μετά να βρείτε τους προδρόμους, να διηλύσετε το υλικό, μετά να το πάτε από την Βραζιλία στη Δυτική Αφρική και από την Δυτική Αφρική να το πάτε στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη στο Αλγεσίρα, σε άλλα λιμάνια και μετά να το διανύμετε. Σε όλα αυτά τα σημεία η αστυνομία μπορεί να σας μαγναρώσει. Στον κυβερνό χώρο όμως μπορείτε να είστε σε αυτό το δωμάτιο και να τα κάνετε όλα αυτά ηλεκτρονικά. Απλώς πρέπει κάπου να μαζέψετε και τα λεφτά. Μόνο εκεί μπορεί να σας πιάσει η αστυνομία. Αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα χωρίς λύσεις και δεν πρέπει να είμαστε εδώ και να θεωρούμε ότι οι εγκληματίες θα καταλάβουν όλο τον κόσμο. Όχι. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Και νομίζω ότι υπάρχουν τέσσερις βασικές ομάδες λύσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να προστατευτούμε στον κυβερνόχωνο. Καταρχήν η συνειδητοποίηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα παιδιά μου ξέρουν τα πάντα για το πώς να κάνουν ποδήλατο, αλλά δεν ξέρουν πώς να αντιδρούν στο διαδίκτυο. Είναι συνέχεια στα κοινωνικά μέσα διαδικτύωσης. έχουν την εμπειρία αυτή. Θα πρέπει να ξέρουν ότι ό,τι βγάζει κανείς στο διαδίκτυο δεν χάνεται ποτέ, δεν θα μπορέσουν ποτέ να το σβήσουν. Πρέπει λοιπόν αυτή η γενιά να μάθει πώς να εμπορεύεται στο διαδίκτυο και πώς να δράσει στο διαδίκτυο. Μετά υπάρχουν οι χώροι προστασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς μια ισχυρή υποδομή για την προστασία αυτή. Αλλά δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό το κυβερνόχωρο. Δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα του εγκλήματος στον πραγματικό κόσμο, κλειδώντας τις πόρτες. Δεν μπορούμε να πούμε στα παιδιά σας μην βγείτε έξω γιατί θα σας επιτεθούν. Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία όπου να μην αποδίδει το κύβερνο έγκλημα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύκολο να αποδώσει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κυβερνοεγκληματίες. Τέλος, χρειαζόμαστε ένα σύστημα διακυβέρνησης του διαδικτύου. Ποιο έχει στην κατοχή του το ίντερνετ. ποιο αποφασίζει αν θα ανοιχνευτούν τα στοιχεία Ποιος αποφασίζει αν κάποιος κλέβει στοιχεία από τα Μητρώα. Κάποιος πρέπει να τα ελέγχει αυτά. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Επομένως, η εντολή για το Ευρωπαϊκό Κέντρο που άνοιξε κυβερνοεγκλήματος που έχει ανοίξει πριν από λίγες εβδομάδες στην Ευρωπόλ. Είναι τα εγκλήματα τα οποία προέρχονται από οργανωμένες ομάδες που οδηγούν σε σοβαρό, σοβαρή ζημιά στα θύματά τους και αυτά τα οποία επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κύριοι στόχοι του EC3. Αυτό το οποίο θέλουμε να είμαστε είναι ένας κόμβος για παροχή πληροφοριών σε σχέση με το κυβερνό έγκλημα, να υπάρχει μια συνολική άποψη για όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι όλες οι χώρες έχουν μια γενικά καλή επισκόπηση, αλλά δεν μπορεί να δει κανείς εάν αυτό το οποίο αντιμετωπίζεται το ερευνάει τη μια άλλη χώρα, γιατί δεν έχουμε ένα κεντρικό, κεντρικό σημείο ανταλλαγή πληροφοριών. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κεντρικό κόμβο που να ανταλλάσσονται πληροφορίε. Μετά πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα εκπαίδευση και δημιουργία ικανότητα, τη λειτουργική υποστήριξη, ή ιατροδικαστική υποστήριξη. Ελπίσουμε με το, τη βοήθεια του προγράμματο Horizon 2020. Αυτό το έγκλημα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσουν μονάχα ιδιοκτικέ δυνάμει. Πρέπει να βοηθήσουμε τις ιδιωτικές, να χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια των ΜΚΟ των ιδιωτικών εταιριών και άλλων φορέων. Επομένω, το να έχουμε επαφή μαζί του είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική και να ελέγχουμε όλα τα μέσα τα ηλεκτρονικά και μαζί με την ίνισα να μπορούμε να προβλέψουμε τι επίκειται. Αυτοί είναι λοιπόν οι χώροι για τους οποίους εμείς θα αναπτύξουμε δραστηριότητα. Θα σταματήσω τώρα εδώ, Κλείνω την παρέμβασή του μου με το να σας ενημερώσω για το πρόγραμμά μας. Πιστεύω από την πρώτη μέρα ότι η δημιουργία του κέντρου για το κυβερνό έγκλημα απαιτεί μια περιεκτική προσέγγιση. Δεν είναι σαν την Ευρωπόλη. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση γιατί έχουμε στο, στην ομάδα μας ένα εκπρόσωπο από την Κομισιόν, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, από την ΕΝΙΣΑ, εγώ, από την ΣΥΠΟΛ, από την Eurojust, από την Ομάδα Δράσης για το Κυβερνό Έγκλημα, για τι ομάδε που αντιμετωπίζουν τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και τέλο από την Πολ. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν αυτό το κέντρο να είναι συμπληρωματικό με το Ευρωπαϊκό Κέντρο. Υπάρχει τόσο πολύ έγκλημα που δεν χρειάζεται να ανταγωνιζόμαστε, υπάρχει για όλους, απλώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους κοινού σπάνιους πόρους μας για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε στη ρίζα το κυβερνοέγκλημα το οποίο αναπτύσσεται και αναδύεται ως λερνέα και ως ύδρα. Πιστεύω ότι έχουμε κάθε δυνατότητα να κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο, αλλά ξεκινήσαμε λίγο καθυστερημένα και έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε για να επιτύχουμε το στόχο μας. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κύβερνο Εγκλήματος θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του μαζί με την ΕΝΙΣΑ ή μαζί με τις ΜΚΟ, τις ιδιωτικές εταιρείες και τα κράτη-μέλη για να κάνει τον κυβερνό χώρο ασφαλή. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Λίγο τρομακτικά αυτά, ε. Αλλά τέλος πάντων, το καλό είναι ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Και είναι θετικό ότι γίνεται πολλή δουλειά όπως φάνηκε και από την παρουσίασή σας. Και έχουμε και άλλη μία παρουσίαση του κύριου Πολ Τίμερς, ο οποίος εκπροσωπεί εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας μιλήσει για το πακέτο που υιοθετήθηκε πρόσφατα όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Ευχαριστώ πολύ. Θα επικεντρωθώ κυρίως σε αυτά που προτείνουμε για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς τα προβλήματα τα οποία ακούσατε μόλις πριν από λίγο όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Υπάρχει λοιπόν μια ε, πρόταση για οδηγία όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Είδαμε πόσο σημαντικός είναι ο ψηφιακό κόσμος για όλους μας σήμερα. Με τη στρατηγική μας λοιπόν προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι θα εξακολουθήσουμε να έχουμε οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό το θέλουμε όλοι. Θέλουμε όλοι να συνεχίσουμε να μπορούμε και να χρησιμοποιούμε και μάλιστα όλο και περισσότερο το διαδίκτυο, αλλά γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία στο επίπεδο της κυβερνοασφάλειας. Υπάρχουν κίνδυνοι, διάφορα συμβάντα έχουν καταγραφεί, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Θέλω όμως να σας πω ότι δεν πρόκειται μόνο για το έγκλημα, μπορεί να είναι και κάτι που απλώς συμβαίνει. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα προέρχεται από αμέλεια ή από ανθρώπινο σφάλμα ή επειδή κάποιος δεν ξέρει πώς να προστατεύσει τον εαυτό του. 9 στα 10 προβλήματα θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί με πάρα πολύ απλούς τρόπους. Είναι θέμα διασυνοριακό βέβαια, θα έλεγα παγκόσμιο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς επικεντρωνόμαστε κυρίως στο τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι και μερικές φορές δεν υπάρχει και αρκετή βούληση για συνεργασία. Προετοιμάσαμε λοιπόν την στρατηγική μας και κυρίως την οδηγία αυτή για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, αφού προηγουμένως είχαμε διαβούλευση με πολλούς φορείς και πολλές συζητήσεις. Αποτέλεσμα των οποίων ήταν ότι 60% των όσων απάντησαν, απάντησαν ότι όντως έχουν ε, βρεθεί αντιμέτωποι με κάποια συμβάντα. Αλλά μόνο το 20% των επιχειρήσεων διαθέτουν ένα σχέδιο διαχείρισης τέτοιων προβλημάτων. Και είναι κρίμα που οι επιχειρήσεις αυτές μάλιστα που ασχολούνται με το εμπόριο αυτό δεν έχουν ένα πραγματικό σχέδιο για να προετοιμαστούν σε περίπτωση που υπάρξουν σχετικά συμβάντα. Πάντως αν κοιτάξουμε γύρω μας, τι βλέπουμε και τι προτείνουμε εμείς δεν έρχεται έτσι κι ε, από τον ουρανό, έχει μια παλιά ιστορία από πίσω του, γιατί έχουν αναλυφθεί μέχρι τώρα διάφορες πρωτοβουλίες η ψηφιακή ατζέντα, για παράδειγμα για την ε, Ευρώπη, η οποία αναφέρεται στο θέμα της ασφάλειας, ε, την προστασία των υποδομών, πολιτική, σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού και ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εκπονηθεί πολλές εκθέσεις και ψηφίσματα τα τελευταία χρόνια. Όλο και πιο πολλά. Και στο Συμβούλιο μάλιστα υπάρχει μια ομάδα η οποία ασχολείται με τον κυβερνοχώρο. Η εικόνα λοιπόν στην οποία καταλήγουμε μας λέει ότι ήρθε πιο καιρός να ασχοληθούμε περισσότερο, να έχουμε μια πιο σφαιρική προσέγγιση και να βάλουμε όλα τα κομμάτια του παζλ μαζί. Και αυτό συμβολίζεται από το γεγονός ότι εκπονήθηκε μία στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια ε, με την βοήθεια της κυρίας Άστον, της Επιτρόπου Μάρστ, που είναι υπεύθυνη για αυτά τα θέματα από τη Γενική Διεύθυνση Home και με την Έλλη Κρούς, την Αντιπρόεδρο, η οποία είναι υπεύθυνη για την ψηφιακή ατζέντα. Φροντίζουν έτσι ώστε και σε επίπεδο υπηρεσιών να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε σε μια στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία. Ε, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Η στρατηγική αυτή τι διασφαλίζει. Τι λέει. Λέει ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να τηρούμε στον κυβερνοχώρο τις αρχές μας, να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας στον κυβερνοχώρο, στον ψηφιακό χώρο και να υπάρχει συγχρόνως σεβασμός και πρόσβαση όλων, αλλά και σεβασμός όλων ε, των αρχών που προστατεύουν τα δεδομένα. Επίσης, η στρατηγική αντιμετωπίζει και τις διάφορες προκλήσεις, την ασφάλεια, την ε, αντοχή. Εδώ, πόσο δηλαδή μπορεί να αντισταθεί το σύστημα αυτό πληροφοριών σε προβλήματα, σε συμβάντα που μπορεί να προκληθούν στο κυβερνοχώρο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το κυβερνοέγκλημα επίσης, ακούσατε μερικά, και πώς θα αναπτύξουμε μια πολιτική σε διεθνές επίπεδα για τον κυβερνοχώρο. Και όλα αυτά, όπως σας είπα πριν, τα αναλαμβάνουν διάφοροι φορείς, διάφορες πλευρές, ιδιωτικός δημόσιος τομέας, οργανώσεις κλπ. Η στρατηγική περιγράφει το ρόλο του κάθε φορέα και σε έναν βαθμό μιλάει και για τη συνεργασία μεταξύ τους και πώς μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία. Πάντως, τη στιγμή τώρα που βρισκόμαστε, τη στρατηγική μας αυτή, την ε, σφαιρική, τη θέλουμε γιατί βάζει διάφορα στοιχεία μαζί, αλλά σε έναν τομέα ο οποίος εξελίσσεται τόσο γρήγορο όπως είναι αυτός, καταλαβαίνετε ότι αυτή η στρατηγική δεν μπορεί να δίνει απάντηση σε όλα. Οπότε είναι μια στρατηγική η οποία θα συνεχίσει να εξελίσσεται θα εξελίσσεται ανάλογα με το τοπίο που διαμορφώνεται, ανάλογα με την εμπειρία που συλλέγουμε και με τη συνεργασία βέβαια των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν ή έχουν κάποια ευθύνη για τη στρατηγική αυτή. Πιο συγκεκριμένα, για να ενισχύσουμε την ε, αντοχή, την αντίσταση δηλαδή των ε, δικτύων και την ασφάλεια θέλουμε να κοιτάξουμε την λυσίδα που προμηθεύει τις προφορίες πρώτα απ' όλα. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας όλα όσα μπορούμε να έχουμε από την έρευνα και την ανάπτυξη. Την συνεργασία ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να αντιμετωπίσουμε τα botnets, όλα αυτά τα συστήματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε κύβερνο επιθέσεις, να ενισχύσουμε την ασφάλεια των συστημάτων επίσης, τα οποία μας προμηθεύουν ενέργεια, ε, ή οτιδήποτε άλλο, τα smart grids που είναι η επόμενη γενιά, και να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση του κόσμου. για το κυβερνό Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος. Συνεργαζόμαστε με την ΕΝΙΣΑ και την Eurogest και ενθαρρύνουμε την ε, ομαλή εφαρμογή της οδηγίας για το κυβερνοέγκλημα. Αυτά περί κυβερνοέγκληματος. Εδώ για την αντίσταση πώς θα γίνεται η ανείχνευση των προγραμμάτων, πώς θα γίνεται η αντίδραση σε αυτά και πώς θα βρίσκουμε μέτρα και λύσεις σε ό,τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί με διάλογο και με συνέργειες. Και ζητάμε φυσικά συνεργασία μεταξύ των χωρών νομελών, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης κλπ. Η στρατηγική αυτή θέλει επίσης μια πολιτική σε διεθνές επίπεδο για τον χώρο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία. Εννοείται ότι από μόνοι μα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι ενδιαφέρον όμω να δούμε ότι μία εβδομάδα μόνο αφού είχαμε την στρατηγική μας αυτή για τον κυβερνοχώρο, ο Ομπάμα επίση έβγαλε ένα, διάκτημα, ένα διάταγμα που αναφερόταν σε αυτό ακριβώ το ζήτημα στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Άρα λοιπόν τι προκλήσει αυτέ θέλουν και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού να τι αντιμετωπίσουν. Θέλουμε επίση να προωθήσουμε το ελεύθερο εμπόριο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η ακρογωνία λύθη αυτή τη στρατηγική μα. Θέλουμε επίση προδιαγραφέ για τη συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο και να στηρίξουμε την ικανότητα, την οικοδόμηση ικανότητας προκειμένου να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν και σε τρίτες χώρες τις προκλήσεις του κυβερνοχώρου. Η οδηγία λοιπόν για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών βασίζεται στο άρθρο 114 της εσωτερικής αγοράς. Και είναι πολύ βασικό αυτό γιατί θέλουμε τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη να τα διατηρήσουμε τη εσωτερική μα αγορά. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Το ένα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, σε εθνικό επίπεδο πρώτα απ' όλα. Χρειαζόμαστε επίση συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ώστε να έχουν τι ίδιε ικανότητε αντίδραση όλες οι χώρες. Γιατί οι συμβάντα μπορεί να συμβούν διασυνοριακά όπως καταλαβαίνετε. Και χρειάζεται επίσης και μια κουλτούρα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κουλτούρα διαχείρισης του κινδύνου και με συνεργασία βέβαια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι κοινέ απαιτήσει τώρα σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μια τέτοια στρατηγική πρέπει να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο πρώτα απ' όλα και να υπάρχει και ένα σχέδιο συνεργασία. Πώ συνεργάζεσαι δηλαδή ο δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα και με τι αρχέ σε περίπτωση κάποιου συμβάντο. Επίση, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να ορίσουν μια αρμόδια εθνική αρχή, ένα κεντρικό σημείο δηλαδή για τη συνεργασία αυτή με τον υπόλοιπο κόσμο. Και βέβαια ναι, έχει, υπάρχει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αντιμετωπιστούν συμβάντα. Αυτό με μια ομάδα που το ονομάζουμε CERT, Computer Emergency Response Team. Η ΕΝΙΣΑ έχει βοηθήσει πάρα πολύ κατά το παρελθόν ακριβώς για να βοηθήσει να δημιουργηθεί αυτού του είδους ικανότητα σε εθνικό επίπεδο και να βοηθήσει να δημιουργηθούν τέτοιες ε, ομάδες αντίδρασης σε περίπτωση συμβάντων στον κυβερνοχώρο. Βασιζόμενοι λοιπόν σε αυτήν την ικανότητα που θέλουμε να αναπτύξουν οι χώρε μέλη σε ικανοποιητικό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχέ μετά πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ του σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουν έγκαιρε προειδοποίησει και να μπορούν συντονισμένα να ανταποκρίνονται σε συμβάντα συμβάντα τα οποία μπορεί να πάρουν τεράστιε διαστάσει πάρα πολύ γρήγορα και ξέρετε πόσο γρήγορα μπορεί να πάρει διάσταση ένα πράγμα στο διαδίκτυο. Και εδώ πρέπει να δούμε και την ευθύνη των ε, χωρών. Δηλαδή πρέπει οι χώρες να ενημερώνουν η μία την άλλη, γιατί πάρα πολύ εύκολα το συμβάν διαχέεται και πάει και σε άλλες χώρες. Και ίσως δεν φτάνει σε μία χώρα να αντιμετωπιστεί το θέμα, ίσως πρέπει να είναι προετοιμασμένες και άλλες χώρες να το αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εμπόριο που είναι διασυνοριακό συχνά. Θέλουμε επίσης, η στρατηγική δηλαδή προβλέπει τα κέντρα κυβερνοχώρου και τακτικές ε, εκθέσεις και αναφορές μεταξύ ομοτήμων. Η Ενίσα βοηθάει σε αυτό. Οι έγκαιρες προειδοποίησεις όσον αφορά τους κινδύνους και τα συμβάντα πρέπει να αναφέρεται και να εντάσσεται μέσα σε γενικότερα σχέδια Αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Έρχομαι τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Πολλοί τομείς μπορεί να βρεθούν ε, θύματα προβλημάτων, οπότε οι αρμόδιε αρχές πρέπει με συντονισμένο τρόπο, όπως είπαμε, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και ποιοι είναι αυτοί οι τομεί, που, για τους οποίους ολοχεύει μεγαλύτερος κίνδυνος, Κάναμε μια έρευνα και είδαμε ότι οι τομείς αυτοί που πρέπει να καλύπτονται από την διαχείριση κινδύνου είναι η ενέργεια, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, τα χρηματιστήρια, οι μεταφορές, αναέριες, θαλάσσιες, σιδηρόδρομοι, υγεία, διαδίκτυο, η πάροχη δηλαδή, και η δημόσια δίκηση. Η προσέγγιση μας βασίζεται στην εμπειρία που έχουμε από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο που ήδη θέτει την ίδια υποχρέωση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Άρα βρισκόμαστε στο ίδιο πνεύμα που βρισκόμαστε και σε άλλους τομείς αλλά τώρα το επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς. Σίγουρα μπορείτε να συζητήσετε, είναι δηλαδή υποσυζήτηση το κατά πόσο αυτοί οι τομείς είναι οι μόνοι. Εμείς καταλήξαμε ότι αυτοί έχουν την μεγαλύτερη σημασία, είναι αυτοί για τους οποίους ελοχεύουν οι περισσότεροι κίνδυνοι, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι. Διαχείριση κινδύνου. Είναι διαφορετικό το επίπεδο ασφάλειας ε, κάθε φορά, οπότε έχει να κάνει με την διαδικασία. Είναι μια δυναμική διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχουν στάνταρτ προδιαγραφές. Ανάλογα με το κίνδυνο και την κατάσταση πραγμάτων λαμβάνονται και τα κατάλληλα μέτρα. Η αναφορά συμβάντων τώρα. Πρόκειται για συμβάντα τα οποία επηρεάζουν τις υπηρεσίες κλειδί στους τομείς που αναφέραμε ώστε να υπάρχουν και εγγύσεις συγχρόνως για τις επιχειρήσεις του απόρριτου δηλαδή ή αν είναι πιο ευάλωτες να φροντίζουμε να λαμβάνουμε και αυτά υπόψη μας. Τώρα, για να επανέλθω στη στρατηγική για την ασφάλεια. Μιλάμε για μια οδηγία, έτσι. Υπάρχει ένα νομοθετικό δηλαδή τμήμα. Αλλά η στρατηγική είναι πιο πλήρης, γιατί περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία, όπως είναι ε, η όθηση της αγοράς, της συνεργασίας δημοσίου ιδιωτικού τομέα, προδιαγραφές, έρευνα, ανάπτυξη. Και βέβαια είμαστε στραμμένοι και στον ορίζοντα του 2020, γιατί φυσικά ο κυβερνοχώρος ε, θα είναι εκεί όλο και περισσότερο σίγουρα θα επηρεάσει πολλούς ε, τομείς καινοτομίε. Μιλάμε σήμερα για συστήματα ευφύους υγείας ή μιλάμε για τις ευφύείς πόλεις και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την αντίσταση σε επιθέσεις ενδεχομένω στον κυβερνοχώρο. Τώρα βρισκόμαστε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο θα μελετήσει την πρόταση αυτή. την οδηγία δηλαδή για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνίων και Ενέργειας ώστε να εξετάσει ολόκληρη αυτή τη στρατηγική. Από εκεί και πέρα και εσείς βέβαια θα εξετάσετε το θέμα και σήμερα περιμένω να έχω αντιδράσεις από σας. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο σε ένα χρόνο να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων συνεχίζοντας με τη στρατηγική αυτή και να έχουμε και μια ετήσια διάσκεψη για το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο υπό τις δύο αντιπροέδρους προκειμένου να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα αυτό που πιστεύουμε ότι είναι ζωτικές σημασίες για την Ευρώπη. Ευχαριστώ, πολύ τους τρεις ομιλητές για τις παρουσιάσεις που ακούσαμε. Ερωτήσεις και απαντήσεις προφανώς. Εκπροσωπούνται εδώ και άλλοι ε, τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα παρά και Συμβούλιο και Επιτροπή. Αν θέλετε πείτε το. Ο πρώτος που ζήτησε το λόγο, ο κύριος Κλέης. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Στον κύριο Πέρς και Έντινγκ. θέλω πιο πολύ να ρωτήσω κάτι. Γιατί αναφέρθηκαν στις μεγάλες απειλές που έχουν ήδη εντοπιστεί για τον κυβερνοχώρο. Και ακούσαμε επίσης ότι είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τους hackers ατομικά, τον καθένα. Ρωτάω λοιπόν, Δεν πρόκειται μόνο όμως για ατομικά ε, δράστες με επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, αλλά υπάρχουν και κράτη τα οποία επιτίθεται στον κυβερνοχώρο. Για την Κίνα ακούσαμε τελευταία ότι συστηματικά και σε μεγάλη κλίμακα μάλιστα ε, παραβιάζει και κάνει και σαμποτάζ ε, κυβερνητικών συστημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, αλλά και στην Ευρώπη σε επιχειρήσεις ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες επιχειρήσεις γενικά. Θα ήθελα λοιπόν από τον κύριο Πάρους ή από τον κύριο Έντινγκ, δεν ξέρω, να ακούσω κάποια απάντηση, δηλαδή τι έχουν να μας πούνε παραπάνω. Δεν θα έπρεπε να μιλήσουμε και για τέτοιες απειλές που προέρχονται από μια χώρα σαν την Κίνα. Καταλαβαίνετε ότι οι εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα ή ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κίνα είναι κάτι που έχει τεράστιες διαστάσεις. Είμαστε έτοιμοι να βρούμε αποδείξεις και να βάλουμε την Κίνα μπροστά στις ευθύνες της. Ευχαριστώ κύριε Κλέης. Κύριε Ιντβέλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους ομιλητές γιατί πολύ, για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Δύσκολο μπορώ να κάνω σχόλια ή να θέσω ερωτήματα γιατί οι τομεί που καλύφθηκαν είναι τόσο εκτεταμένοι που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλάμε πια. Χρειάζονται μέτρα σε τομείς από όπως που ξεκινούν από την εσωτερική αγορά, την ασφάλεια, την άμυνα. Μιλάμε για τομείς τελείως διαφορετικούς όπου η Ένωση έχει τελείως ε, διαφορετικού επίπεδου εξουσίες. Η αστυνόμευση στον κανονικό κόσμο είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την άμυνα. Υπάρχουν άλλα επίπεδα ασφαλείας ε, για τις πολιτικές ελευθερίες. Βλέποντας μια διαφάνεια που λέει για ακτιβισμό ή ακτιβισμό τρομοκρατία, ανησυχώ. Μπορεί να μου πείτε πώς διακρίνουμε. Ε, ε, οι γραμμές μεταξύ των θέσεων είναι πολύ φλού. Μιλάτε για απάτη, μιλάτε για παράνομη, παράνομο κατέβασμα που είναι, βία, που είναι παραβίαση του copyright, σεξουαλική εκμετάλλευση του μέχρι στρατιωτικέ επιθέσεις και τρομοκρατία. Είναι διαφορετικοί τομείς. Εγώ είμαι υπέρ της διεπιστημονικής συνεργασίας, αλλά παρά είναι μεγάλο. Ρίχνουμε τα πάντα σε ένα καλάθι, μόνο και μόνο γιατί γίνεται στο ίντερνετ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό κριτήριο στο οποίο πρέπει να βασίσουμε την πολιτική μας. Αν ακούω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, αν ακούσω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα για παράδειγμα που περιλαμβάνει εκπροσώπους της, εξωτερι... της εξωτερικών σχέσεων. Μπορεί να μας εξηγήσετε πώς ενεπλάξαν αυτοί σε αστυνομική δομή. Επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το είδος των πολιτικών που συζητούμε, τις εξουσίες που δίνονται, τις εγγυήσει που υπάρχουν και τους στόχους που επιδιέκονται. Μετά υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Τέθηκαν ερωτήσεις για άλλες χώρες κυβερνήσεις, έθνη που μπορεί να επιτίθεται σε συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις, πρόσφα... τις τελευταίες μέρες ακούσαμε πληροφορίες για κατηγορία επίθεσης που οργάνωσε η κινησική κυβέρνηση σε αμερικανικές υποδομές. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το εντοπίσει αλλά νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον να ρωτήσουμε εμείς τι κάνουμε, οι κυβερνήσεις Ένωσης τι κάνουν. Λέμε να προστατεύουμε τα συμφέροντα της Ένωσης από τις εξωτερικές επιθέσεις και αν υπάρχει εμπλοκή της υπηρεσία εξωτερικής δράσης αυτό σημαίνει ότι και εμείς θα κάνουμε τέτοιες επιθέσεις, οικονομικές επιθέσεις και αν ναι θα το αποφασίσει. spying illegally. Uh, και μετά, άλλο ερώτημα. Κυβερνήσεις της Ένωσης που παρακολουθούν τους πολίτες της, δεν ξέρω την ορολογία, το ξέρει ο Γιάνν Άλμπερτς ε, περισσότερο, αλλά θυμάμαι ότι οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της ε, Ολλανδίας αγόρασαν παράνομο spyware για να χρησιμοποιήσουν κατά των πολιτών τους. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες πρέπει να συμπεριλάβουμε στην προστασία και την προστασία των πολιτών από τις κυβερνήσεις τους. Η κυρία Ζίμπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά που ακούσαμε σήμερα δεν νομίζω ότι ήταν αναλυθή αλλά αναρωτιέμαι τι καινούριο είχαν όλα αυτά ότι κάποιος πόλεμος λαμβάνει χώρα ουσιαστικά στο κυβερνόχωρο. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό τουλάχιστον εδώ και 10-20 χρόνια το ξέρουμε. Έχουμε συνέχεια εκθέσεις που μας λένε πόσο αδύναμοι και απροφύλακτοι είμαστε σε αυτό το κυβερνόχωρο, σαν άτομα, σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σαν ε, ε κυβερνητικοί οργανισμοί, σαν ε, εργοστάσια, σαν νοσοκομεία πόσο εύκολο είναι κάποιος να μπει και να πάρει τα δεδομένα ή να κάνει δολιοφθορές εκεί. Αναρωτιέμαι. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην ε, Ευρώπη είναι κάτι το οποίο πρέπει να δίνει λαβή σε τόσο ακριβές αναλύσεις και σταθερούς μηχανισμούς αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος. Όταν είναι τόσο εύκολο να υπάρξει παρίσφρηση σε συστήματα υπολογιστών. Μιλάμε για θέματα όπως είναι η ασφάλεια των δεδομένων, η αρμοδιότητα των μέσων ενημέρωσης και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα τα οποία είναι πιο σημαντικά για μένα να είναι η εστίαση της προσπάθειάς σας από αυτά τα οποία είπατε, γιατί εκεί υπάρχει πράγματι η δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν συνέχεια εκθέσεις για το πώς γίνεται το hacking. Αλλά μπορεί να σας φαίνεται κοινικό αυτό που λέω, αλλά είναι περιορισμένης κλίμακος αυτό. Αλλά τα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά είναι να αντιμετωπίσουμε πιο ουσιαστικές απειλές. Δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος προσπάθησε να γονατίσει όλη την ηλεκτροπαραγωγή στις χώρες μας. Είναι πιο σημαντικό λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πιο σημαντικά προβλήματα και όχι να ξοδεύουμε εκατομμύρια για θέματα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα με ένα κεντρικό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθηθούν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα πρώτο σχόλιο, γιατί αυτό νομίζω ότι αναφέρθηκε στην πρώτη παρέμβαση. Ε, των ομιλητών. Δεν νομίζω ότι οι hackers είναι γενικά εγκληματίες. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν οι hackers οι οποίοι υποδείκνυαν τα ασφάλματα και τα κενά ασφαλείας και βοηθούσαν τις επιχειρήσεις και τους άλλους χρήστες να κλείνουν τις τρύπες όταν οι κυβερνήσει δεν κάναν τίποτα για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει λοιπόν να κατηγορήσουμε αυτού οι οποίοι μα έχουν αποκαλύψει τα προβλήματα ασφαλεία και σίγουρα δεν πρέπει να του αποκαλούμε εγκληματίε. Προφανώ υπάρχουν και εγκληματίε οι οποίοι προσπαθούν να παραβιάσουν τα συστήματα ασφαλεία και τα συστήματα προστασία των υποδομών. Όπω είπα προηγουμένω και την προηγούμενη φορά, εγώ υποστηρίζω το να δημιουργηθεί τη δημιουργία του κέντρου για το κυβερνό έγκλημα της Europol είναι χρήσιμο να υπάρξουν περαιτέρω έρευνα, έρευνες για τα κενά ασφαλείας τα οποία υπάρχουν στα δίκτυα και που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα. Όταν βλέπω όμως την προτινόμενη οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και της πληροφορίας, έχω να κάνω κάποια σχόλια. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να μας απασχολεί μονάχα η ανακοίνωση των παραβιάσεων σε περιπτώσεις που έχει γίνει ήδη η ζημιά. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας ε, απασχολήσουν και τα τροτά σημεία εκεί που υπάρχουν κενά ασφαλείας, όπου δεν υπάρχει πραγματική αντίληψη ασφαλείας και δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα για την αντιμετωπίση αυτή. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε κάτι και για την αστική ευθύνη της μη εφαρμογής συστημάτων ε, ασφάλειας. Μπορούμε εδώ να συζητήσουμε και με την Ενίσα για τα εργαλεία τα οποία είναι πιο πρόσφορα για αυτό το στόχο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να εστιάσουμε μόνο σε αυτούς οι οποίοι διατηρούν τις πληροφορικές υποδομές. Υπάρχουν πολλά συστήματα που δεν έχουν μόνο το χαρακτήρα κλασικών υποδομών, αλλά είναι και συστήματα που πρέπει να έχουν τα δικά τους συστήματα ασφαλείας. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε σχέση με τις προτάσεις αυτές, αλλά και αυτό είναι το τελικό μου σχόλιο. Θα ήθελα να, συνεχίσω, να αυτό που ξεκίνησε να λέει η Σοφή Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να τα βάλουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Θα ήθελα να εστιάσουμε στα σημεία αυτά όπου υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα και εκεί θα πρέπει να το λύσουμε με πρακτικά μέσα, με τα κατάλληλα ε, μέσα αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι σκόπιμη η συζήτηση αυτή για την εγκληματικότητα και την ασφάλεια στον χώρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πούς ε, και τον κύριο Τρόις καθώς και τον κύριο Τίμερς για την συνεισφορά τους. Ωστόσο, έχω ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια είναι ανάγκη και προφανές όμως έχουμε σίγουρα να κάνουμε με ένα εγκάρσιο και διεπιστημονικό θέμα. Επηρεάζει στην ίδια την Επιτροπή, την κυρία Κρούς, την κυρία Άστον, την κυρία Μάρτστον. Ταυτόχρονα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο τομέα, την κυβερνοασφάλεια, την κυβερνοεγκληματικότητα, την κυβερνοάμυνα αφετέρου τονίζεται ότι χρειάζεται μια κοινή αρχή, δηλώνεται ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει μια ετήσια διάσκεψη, ένα χρονοδιάγραμμα. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά. Και είναι μια ερώτηση που απευθύνω προς τον κύριο Τίμερς. Είπατε, κύριε Τίμερς, πολλές φορές στην παρέμβασή σας, ότι πρέπει να, πρέπει να, πρέπει να, υλφώ. ρωτώ, για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πρέπει, τι λεφτά έχετε, ποια είναι η κάλυψη του προπολογισμού. Δεν έχει νόημα να μας δίνετε στόχους που συνδέονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική που σίγουρα είναι απαραίτητη και απαράγραπτη, αλλά τζάπα. Παρουσιάζεται δηλαδή σε 7 Φεβρουαρίου μια στρατηγική τι χρήματα δώσατε ή απλά έχουμε μια πανέμορφη δήλωση προθέσεων με συζήτηση που δεν γίνεται. Η Europol έχει προϋπολογισμό έξτρα για αυτή τη νέα δραστηριότητα. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την Europol, για τα υπόλοιπα το ίδιο είναι. Ευχαριστώ. Μωράες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τους ομιλητές, όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Η ερώτησή μου αφορά τον κύριο Τίμερς. Κατανοώ απόλυτα αυτά που λέει η κυρία Ιντενβερτ για το ότι μας δώσατε ένα τεράστιο πλέγμα θεμάτων. Όταν υποβλήθηκε το πακέτο στο ξεκίνημα του Φεβρουαρίου από την κυρία Κρούση και την κυρία Άστον, το πρόβλημα που είχαμε στο Κοινοβούλιο ήταν ποιος είναι ο υπεύθυνος. Στις Ηνωμένε Πολιτείες ένα από τα βασικά εργαλεία που έχει οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, είναι ότι ο πρόεδρος Ομπάμα έβγαλε μια, ένα διάταγμα που αντιμετωπίζει το έγκλημα. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Η ερώτηση είναι προς τον κύριο Τίμες. Αυτό το κάνουν ούτως ή άλλως τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι στο ξεκίνημα στην παρουσίαση ε, που έκανε η κυρία Κρός είπε ότι πολλά από τα κράτη-μέλη δεν λειτουργούν επαρκώς στον τομέα αυτό που ήδη μας ανησυχεί τι είναι ενδεδειγμένο κατάλληλο να γίνεται στο θέμα του κυβερνού εγκλήματος. Ο κ. Άλμπερτ ανέφερε ότι όταν σε 7 Φεβρουαρίου έγινε η παρουσίαση, ε, στο δικό μου κράτος ε, οι πληροφορίες ήταν για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων να αναφέρουν τις περιπτώσεις hacking. Αυτό είναι σημαντική απέτηση να υπάρχει δηλαδή αναφορά του κυβερνού εγκλήματος. πιο σημαντικό είναι να παρουσιάζονται οι αδυναμίες στο σύστημα. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, στο πακέτο αντιμετωπίζουμε αυτό που θεωρεί ο κόσμος ως το μεγάλο κυβερνό έγκριμα. Έγινε ανάλυση στα κράτη-μέλη. Τι πρέπει να κάνουμε σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο ούτω ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη από πλευρά κόσμου. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Κατόπιν είδαμε να, κατά πόσο υπάρχουν προβλήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων μεταξύ αυτού και του πακέτου προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όλοι λέμε ναι, αλλά α δούμε και τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα πριν ξεκινήσουμε με κάτι προφανέ ε, που όλοι το θέλουν αλλά που δημιουργεί προβλήματα από την οπτική γωνία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρία Φαγιών, Ευχαριστώ τους ομιλητές. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπαν. Στο παρελθόν πολλές φορές ακούσαμε το κίνδυνο που υπάρχει για το ίντερνετ, από το ίντερνετ. Όντως φοβίζει και δεν έχω συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις. Σήμερα το πρωί είχα και ένα ενδιαφέρον πρωινό για το κυβερνοέγκλημα με κάποιους εμπειρογνώμονες. Το θέμα είναι ότι δεν είναι εθνικό, αλλά διασυνοριακό έγκλημα. Ξέρουμε ότι πολλά λεφτά παίζονται στο ίντερνετ, κυκλοφορούν μέσω του ίντερνετ. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι πολλές επιχειρήσεις ε, χάνουν εμπορικά ε, μυστικά, δηλαδή τις πληροφορίες που έχουν από πατέντες ή από την εκμετάλλευση συγκεκριμένων Έχουμε, άλλοι αναφέρουν ότι υπάρχει ένα πολύ κατακαιρματισμένο νομικό πλαίσιο κατά του εμπορικού, κατά του εγκλήματος. Χρειάζεται καλύτερος έλεγχος του πού πηγαίνουν τα χρήματα. Ερώτηση, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε οργανωμένο έγκλημα, super hackers. Δεν μπορούμε να τους βρούμε. Πώς θα χτυπήσουμε το έγκλημα αυτό. Υπάρχει τώρα ένα κέντρο κυβερνοεγκλήματος και για σας ε, απευθύνεται ερώτηση κύριε Έτινγκ, εσείς ξεκινήσατε πρόσφατα. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει τέτοια δυνατότητα σε όλα τα κράτη-μέλη. Πώς είναι η συνεργασία, πώς μπορείτε να πετύχετε Μπορούν τα κράτη-μέλη να παρέμβουν εκ των προτέρων στο κέντρο. Τι κάνετε για να κάνετε ανταλλαγέ πληροφοριών μεταξύ αστυνομία, δικαστηρίων, εισαγγελία. Πώς μπορείτε να προχωρήσετε περαιτέρω. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό καθεστώς, συστηματικότερους ελέγχους και δεν ξέρω πώς να προχωρήσουμε στο Κοινοβούλιο ενώ θα είμαστε συνεχώς ένα βήμα πίσω. Είπατε κι εσείς κύριε Πέσσερ ότι το μέλλον είναι σαν ένα μετεωρολογικό δελτίο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φαγιάννη. Πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσεις. Απαντήσει τώρα. Δεν ξέρω, είναι εδώ τα άλλα θεσμικά όργανα, η Επιτροπή, το Συμβούλιο, μήπως ε, θέλουν να παρέμβουν. Όχι. Ωραία, απαντήσει τότε. Δεν είναι εδώ Επιτροπή Συμβούλιο, δεν θέλουν τίποτα έτσι. Όχι. Καλώς. Με την ίδια σειρά. απαντήστε στα σχόλια και στις ερωτήσεις, παρακαλώ. Ο κύριος Πέρσερ πρώτα. Παρακαλώ κύριε Πέρσερ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσε οι ερωτήσεις, πράγματι. Θα προσπαθήσω με τη σειρά να τις απαντήσω. Η πρώτη είχε, κάνει, είχε να κάνει με την ευθύνη χωρών ε, για, τα, για Εντάξει, υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν τα ίχνη στο διαδίκτυο και ακόμα και οι πιο ειδικοί δεν καταφέρνουν να βρουν από πού ακριβώς προέρχονται επιθέσεις. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι όμως δικιά μας εντολή αυτό εμείς. Αντί να ψάξουμε να βρούμε ποιος κάνει την επίθεση, προσπαθούμε να βρούμε πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για να σταματάμε τις επιθέσεις, για να μην γίνονται σε εμά. Ο ο ιδιωτικό, ο δημόσιο τομέα, ε, οι χώρε να είναι προετοιμασμένοι όσο γίνεται καλύτερα από όπου και αν προέρχονται επιθέσει. Δηλαδή, καλό αυτό που λέτε, αλλά ξέρω ότι σα απογοητεύω με την απάντησή μου. σω ε, ο συνάδελφο να μπορεί να σα βοηθήσει περισσότερο. Τώρα, αναφερθήκαμε στις απειλές. Ευθύ εξ αρχή. Πολλοί είπαν ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Εντάξει, δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν είμαστε και σε καταστροφική κατάσταση. Εκατομμύρια επιθέσει λαμβάνουν χώρα συνέχεια. Στον χρηματοοικονομικό τομέα, για παράδειγμα, που ξέρω εγώ, συνέχεια γίνονται. Συνεχώ. Στην Ευρώπη τα καταφέρνουμε αρκετά καλά γιατί τελικά δεν έχουμε τόσο πολλές περιπτώσεις με μεγάλη ζημιά. Έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο ρημότητας, δηλαδή χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειες. Όχι, και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί έτσι κι αλλιώς. Όσο καλή και αν γίνουμε στην αντιμετώπιση, στην πρόληψη, ο αντίπαλος θα προσαρμοστεί και θα βρει νέες μεθόδους. Άρα συνέχεια θα πρέπει να προσπαθούμε και θα επανέλθω και αργότερα. Η προστασία δεδομένων. Είπατε ότι δεν θα πρέπει όλα να τα βάζουμε στο ίδιο καλάθι και δεν το κάνουμε. Η νομοθεσία είναι διαφορετική στην πολιτική αντιμετώπιση των εγκλημάτων, αλλά πρέπει παράλληλα να τα βλέπουμε όλα, γιατί αποτελούν τις δύο του ίδιου νομίσματος. Χρειαζόμαστε καλή ασφάλεια για να προστατεύουμε και χρειαζόμαστε προστασία των δεδομένων άμα θέλουμε να έχουμε καλή ασφάλεια. Και τα δύο χρειάζονται δηλαδή και τα δύο πρέπει να τα έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Δεν μπορεί να έχεις ε, εξαίρετη προστασία δεδομένων και εξαίρετη ασφάλεια. Άμα θέλεις να προσέξεις την ασφάλεια μπορεί να πρέπει να ασχοληθείς και με τα προσωπικά δεδομένα. Οπότε τι λέμε, λέμε ότι η έλεγχη είναι αρκετά καλή, ε, γίνονται με υπεύθυνο τρόπο ότι υπάρχει καλή ισορροπία ανάμεσα στην προσπάθεια να πιάσουμε τον κακό και από την άλλη μεριά να προστατεύουμε και τα προσωπικά δεδομένα. Έγιναν ε, κάποιες, ε, ε, κάποια σχόλια για τον πόλεμο στον κυβερνοχώρο και πόσο προετοιμασμένοι είμαστε. Σας είπα ότι είμαστε αρκετά καλά προστατευμένοι, αλλά μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Σημασία έχει πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματά μας. Έχουμε διάφορα μέσα στη διαθέσή μας. Το κέντρο για το κυβερνοέγκλημα είναι ένα, η ΕΝΙΣΑ είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Δεν πρέπει να υπάρχει πολύ κατακαιρματισμένη διαδικασία. Δεν θα πρέπει δηλαδή να φτιάχνουμε καινούρια όργανα συνεχώς. Ξέρω ότι η ΕΝΙΣΑ ξοδεύει πάρα πολύ χρόνο για να ευθυγραμμίσει τις προσπάθειες και να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, αντί να προσπαθούμε να βρούμε άλλα και να ξοδεύουμε έτσι χρήματα χωρίς λόγο. Το θέμα του πόσο τρωτοί είμαστε και αν το κοιτάμε αρκετά, το κοιτάμε. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά για να ξέρουμε πόσο ευάλωτοι είμαστε και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Και να σας πω και κάτι που μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά το ξέρω από πρώτο χέρι. Αν έχετε μια λύση για να μην είσαστε ευάλωτοι, δεν μπορείτε πάντα να τη χρησιμοποιήσετε. Μερικές φορές η λύση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ότι το γεγονός ότι είσαστε ευάλωτοι. Γιατί λύσεις μπορείτε να βρείτε για ένα εύρος υπηρεσιών ή συστημάτων. Πριν από 15 χρόνια, εγώ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανέπτυξα ένα σύστημα που ήταν ε, για να μπορεί να έχει κανείς εμπιστοσύνη στο κομπιούτερ του. Ήταν ένα σύστημα από τις Ηνωμένε Πολιτείες με συγκεκριμένα κριτήρια. Πέρασαμε πολύ χρόνο να το αναπτύξουμε και όταν τελικά φτάσαμε στην εφαρμογή δεν λειτουργούσε. Και γιατί, γιατί οι εφαρμογές είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τον παράγοντα του τροτού χαρακτήρα. Οπότε εντοπίζουμε μεν τον τροτό χαρακτήρα, αλλά να ξέρετε ότι περισσότερο έχει σημασία να προσέξουμε τον μελλοντικό σχεδιασμό, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα και μετά να αντιμετωπίσουμε ε, τα τροτά σημεία τα οποία θα παραμείνουν βέβαια για λίγο καιρό. Μιλήσατε επίσης ε, για το πολυδιάστατο του κυβέρνου εγκλήματος. Ε, πράγματι, γι' αυτό και δεν θέλουμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Πρέπει να χωρίζουμε ότι μπορεί να χωριστεί, αλλά να κάνουμε κοινή ανάλυση όπου πρέπει να γίνει κοινή ανάλυση. Νομίζω ότι προχωράμε βάσει ενός καλού συμβιβασμού. Η νέα στρατηγική και οδηγία είναι κάτι πολύ καλό. Αν κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε νομίζω. Εκεί που μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, ναι, υπάρχει ζήτημα με τον προπολογισμό, με τους πόρους και αυτό μπορείτε να το αλλάξετε. Είμαστε βέβαια εν μέσω οικονομικής κρίσης. Όλοι λένε ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα και το κάνουμε. Αλλά όσο ξαπλώνονται περισσότερο οι απειλές και το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο μεγάλο, εννοείται ότι πρέπει να βάλουμε περισσότερα χρήματα για να διατηρήσουμε την ισορροπία. Όχι για να φτάσουμε στα άκρα και να γίνουμε βασιλικότερο του βασιλέως, όχι, αλλά προκειμένου να διατηρήσουμε την ισορροπία. Πρέπει να επενδύουμε θεμελιώδη δικαιώματα. Το προσέχουμε συνεχώς. φροντίζουμε ό,τι κάνουμε να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το ξέρω ότι ισχύει και για τους συναδέρφους μου. μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμα καλύτερο. Εννοείται, θα χρειαστεί όμως χρόνος. Οι διαδικασίες εξελίσσονται έτσι κι αλλιώς. Και οι χώρες δεν είναι ακόμα σε θέση να κάνουν τα πάντα. Το καλό όμως είναι ότι δουλεύουμε πάνω στην υπόθεση αυτή. Τώρα ότι υπάρχουν super hackers που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Ε, ναι, όντως, δεν υπάρχει τίποτα καινούριο εδώ, αλλά δεν είναι και ανησυχητικό. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε όλους. Ποτέ δεν θα μπορούμε όλους να τους εντοπίσουμε, γιατί και οι δράστες βρίσκουν καινούρια κόλπα. Η ισορροπία είναι αυτό που μετράει. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο δείχνουν. Ναι, θέλουμε περισσότερο προπολογισμό, περισσότερους πόρους. Πάντως, η στρατηγική για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος είναι θετική, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, ας την ακολουθήσουμε και θα δούμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Έρτινγκ, η σειρά εγώ θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε ο Στιβ Πούρσε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στρατηγική για τον κυβερνόχωρο. Είναι μια σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι είναι εξισορροπημένη. Δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες γιατί αυτό δεν είναι μέσα στην ε, αρμοδιότητά μας. Εμείς κοιτάμε την αγκληματικότητα. Απλώς παρακολουθούμε επιθέσεις αυτού του είδους γιατί το πρόβλημα στο διαδίκτυο είναι ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιείτε είναι ακριβώς οι ίδιες. Είτε κλέβετε πληροφορίες, είτε κλέβετε λεφτά. Δεν είναι εύκολο να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος των hackers, γι' αυτό πρέπει να δούμε τι κάνουν. Κυρία Ένφελτ, εγώ κατανοώ ότι είναι πολλά πράγματα που τα βάζουμε στο ίδιο καλάθι και ίσως είναι υπερβολικό. Και στέκομαι στο κυβερνό έγκλημα υπάρχουν μερικές φορές φαιές περιοχές. Και μπορεί κανείς να πρέπει να μπει σε τομείς που δεν είναι ο δικός του τομέας. Και θα πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν ορισμένε τεχνικές οι εγκληματίες. Μπορεί να δουλεύει κανείς για μια κρατική δομή, για μια οργάνωση. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία από πού προέρχεται κανείς. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι παρίσφυσης. Εγώ θέλω να παραμείνω στον χώρο του εγκλήματος αυτή είναι η εντολή μας. Δεν θα κάνουμε τίποτα περαιτέρω αυτού, αλλά πολλές φορές υπάρχει και μια θεά περιοχή πρέπει να λάβουμε υπόψη. Λέτε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης. Βγάλανε <clears throat> το θέμα της δημιουργίας ικανότητας έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς κάνουμε μια αξιολόγηση κινδύνου για τις ε, πηγές κινδύνου που και περιοχές έξω Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούν μετά αυτήν την αξιολόγηση για να δούνε πού πρέπει να γίνει η οικοδόμηση ικανότητος. Υπήρξε και το άλλο ερώτημα, τι κάνουμε για να βοηθήσουμε τις μικρές εταιρείες για να είναι ασφαλείς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ανέφερε και ο Στίβ. Θέλουμε να αυξήσουμε την προστασία και θα ζητήσουμε από τα κρατη να έχουν πιο έντονες διοκτικές δραστηριότητες και να τους εμποδίσουμε από το να καταστρέφουν τις πληροφορίες των επιχειρήσεων. Από τον κύριο Άλμπερτ υπήρξε αυτή η διάκριση μεταξύ καλών και κακών χάκες που κάποιοι είναι κακοί και κάποιοι είναι καλοί. Εγώ ω δημόσιο υπάλληλο δεν μπορώ να έχω μια πολυτέλεια τέτοια άποψη. Εμεί απλώ υποστηρίζουμε τα κρατημέλη γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, δεν κάνουμε εμεί τι δικέ μα έρευνε, έρχονται από τα κρατημέλη. Οτιδήποτε είναι παράνομο, ζητούμε να εφαρμοστεί γι' αυτό η νομοθεσία. Πρέπει να τονίσω επίσης ότι έχουμε ένα πάρα πολύ αυστηρό καθεστώς προστασίας δεδομένων στην Ευρωπόλ δεν θέλω να αναφερθώ στο δικό μου κράτος, αλλά είναι πιο υψηλό το επίπεδο ασφάλειας στη Europol από ότι είναι στη δική μου χώρα. Δεν απελευθερώνουμε ποτέ δεδομένα εάν δεν τα έχουμε ελέγξει. Εμείς περιμένουμε να πάρουμε άλλους 10 ελεγκτές από την κοινή μονάδα για τον έλεγχο των δεδομένων, επομένω υπάρχει πάντα έλεγχος για όλα αυτά. Ο κύριο Ντίμερα ρώτησε αν έχουμε λεφτά. Όχι, είναι άδειε οι τσέπε μας στην ε, Europol δεν έχουμε για το 2013 καμία δυνατότητα. Τα χρήματα που χρησιμοποιούμε για το κέντρο κυβερνοχώρου βγαίνουν από τον ε, τωρινό μας προϋπολογισμό και άλλες περιοχές περιορίζονται για να μπορέσουμε να παίξουμε ένα σοβαρό ρόλο στον τομέα αυτό. Αλλά από ό,τι ξέρω, στο προϋπολογισμό του 2014 θα είναι το τέλος του, της σύραγγος και ελπίζω ότι θα γίνει πραγματικότητα. Κυρία Φαγιών. Έχουμε καλούς εγκληματίες, βεβαίως, έχετε μεγάλο δίκιο. Αυτοί που μπαίνουν φυλακή είναι μάλλον οι χαζοί. Οι ξύπνοι είναι έξω. Και αυτό αφορά και το κανονικό έγκλημα και το κυβερνό έγκλημα. Και μάλλον θα εξακολουθήσει να είναι έτσι. Πρέπει όμως να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας και συμφωνώ με τον Στίβο ότι κάπως τα καταφέρουμε κιόλα. Πρέπει να κατανοήσετε ότι πολλές οργανώσεις αστυνομικές δημιουργούν ικανότητα χωρίς να έχουν και χρήματα. Επειδή ασχολούμαστε με το κυβέρνο έγκλημα, δεν σημαίνει ότι ασχολούμαστε με το κανονικό έγκλημα. Και όταν υπάρχει λιτότητα στον προϋπολογισμό, θεωρούν ορισμένοι ότι αν έχετε υψηλό επίπεδο απασχόλησης, υπάρχει μεγάλο, αν υπάρχει μεγάλο επίθεμα επίπεδο ανεργίας, έχετε και μεγάλη εγκληματικότητα. Αυτό το έχουμε δει στο διαδίκτυο. Υπάρχουν χώρες που έχουν καλά συστήματα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία κτλ. Πρέπει να βοηθήσουμε όμως σε άλλες χώρες που δεν έχουν τόσο καλό σύστημα να υπάρξει αυτή η αλληλεγγύη για να βοηθήσουμε αυτά τα κράτη γιατί όλοι πρέπει να είμαστε ισχυροί και πιο ισχυροί από το πιο αδυνατό κρίκο. Έχουμε προβλήματα με τους ε, hackers οι οποίοι χρησιμοποιούν τις τρύπες που ξέρουν που μπορούν να κλέψουν λεφτά. Επίσης μπορεί να υπάρξει πειρατεία στον υπολογιστή σας και να μην μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. 3% από τους υπολογιστές οι οποίοι έχουν μολυνθεί από ιούς τελικά είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν. Οι τρόες για τις τράπεζες είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε γιατί οι τράπεζες απλώς πληρώνουν και δεν λένε τίποτα. Στις απάτες για τις πιστοτικές κάρτες όταν δεν υπάρχει κάρτα 60% όλων των περιπτώσεων 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο χάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 65% γίνονται χωρίς να έχει ο hacker την ε, πιστοτική κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει αυτά τα συστήματα να γίνουν πιο ασφαλή και το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα πληρωμής με κινητό και αυτά τα συστήματα που γίνονται με Bluetooth στο Starbucks και σε άλλα καταστήματα. Εμείς ήδη ασχολούμαστε και με άλλα θέματα. Η Eurojust έχει ένα σύνδεσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως ακολουθούμε αυτές τις περιπτώσεις και προχωρούμε σε δίωξη. Θα έχουμε συζητήσει και με την Ενίσσα αν μπορούμε να έχουμε σύνδεση και με άλλους φορείς και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερη συνεργασία και η αστυνομία είναι πολύ πιο θετική στο έγκλημα από ότι στο κανονικό έγκλημα γιατί εκεί προστατεύουν ίσω περισσότερο τι πληροφορίε του, αλλά για το κυβερνοέγκλημα διαμοιράζονται περισσότερο τι πληροφορίε που έχουν. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε και είναι ανηφόρα, αλλά θα φτάσουμε. Ευχαριστώ. Ο, κύριο Τίμερ. Ομαδικά θα απαντήσω σε κάποιες ε, ερωτήσει. Πρώτον, ποια είναι η ανάλυση μα, ε, τι θέλουμε να πετύχουμε και από πού ξεκινάμε. π.χ. τι γίνεται επί τόπου. Ακούσαμε ότι κάποια από τα στοιχεία ανάλυση της ΕΝΙΣΑ και της Europol. Ακούσαμε την ανάλυση για το βαθμό προπαρασκευή, το έφεσε ο κύριος Μωράες, την ανάλυση για την ε, ετοιμότητα των κρατών μελών, αλλά και του ιδιωτικού τομέα και των καταναλωτών. Κάναμε πολλές αναλύσεις, αφρίζοντα ε, στοιχεία από διάφορες μελέτες, εκθέσεις κλπ. Πολλά περιλαμβάνονται στον, στην έκθεση αντίκτυπου κινδύνου. Αυτό έγινε σε δύο, γίνεται σε δύο φάσεις. Πρώτα ρωτάμε τα κράτη-μέλη πόσο έχετε προχωρήσει, έχετε ένα πρόγραμμα συνεργασίας για να αντιμετωπίσετε τέτοια επεισόδια και βλέπετε πώς τα κράτη-μέλη ομαδοποιούνται βάσει της ετοιμότητάς τους στην Ευρώπη. Αυτό το βρίσκεται στη σελίδα 23 της, του αντίκτυπου κίνδυνου. Προφανώς αλλάζει αυτό, αλλά είναι και κομμάτι των input. Ένα σημαντικό θέμα είναι ότι δεν έχουμε και επαρκή πληροφόρηση. Πόσο είναι το κόστος ακριβώς των επεισοδίων; Θα βρείτε στοιχεία που αποκλίνουν. Άκουσα 100 δισεκατομμύρια. Άλλοι είπαν για 750 δις. Τα, τα τα συμβάντα σε επιχειρήσεις είναι από 1 έως 60 εκατομμύρια. Όλα αυτά σχετίζονται με την ανάλυση και την παρουσίαση εκθέσεων. Τι θέλουμε να πετύχουμε τώρα. Είδαμε ότι τα προβλήματα αυτά είναι, συνδέονται μεταξύ τους και δεν πρέπει να τα βλέπουμε με μια υπερβολικά μειοπική προσέγγιση. Χρειάζεται να μπορούμε να αφρίζουμε στοιχεία Είχαμε προσεγγίσει σε πολλούς τομείς, αλλά ανεπαρκής. Υπήρχε ένα ανεπαρκές επίπεδο προετοιμασίας και ανεπαρκής ικανότητα αντίδρασης στα κύβερνα επεισόδια. Συνολικά, ο στόχος της στρατηγικής διατυπώνεται ως προς το ότι η Ένωση θα έπρεπε να παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία και ασφάλεια με ένα ασφαλές σύστημα online. Τώρα, είναι πάρα πολλά μαζί. Όχι. Αυτό νομίζω απαιτείται αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν οι διάφοροι φορείς και παράγοντες να μετάσχουν σε μια κοινή στρατηγική. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει focus. Έχουμε το στόχο, έχουμε την ανάλυση, αλλά πρέπει να προχωρούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Σα έδειξα ένα παράδειγμα, την πρόταση της οδηγίας που είναι σαφής για το τι θέλουμε Αυτό που μπορεί να θέσετε είναι πώς αντιμετωπίζεις το interface μεταξύ των διαφόρων τομέων. Ανθεκτικότητα, έγκλημα, διεθνής πολιτική. Αυτό ορίζεται ρητά στην οδηγία και το interface μεταξύ των τομέων ανθεκτικότητας και εγκλήματος σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεις ότι υπάρχει έτοιμα, ζητείτε να υπάρχει συνεργασία. Σε άλλες περιπτώσεις δίνουμε τις υποστηρικτικές δράσεις για το σκοπέ αυτό. Μια πλατφόρμα για παράδειγμα που θα βοηθήσει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που είναι ανεπαρκής δημιουργώντας πρακτικές και διαδικασίες που εν τέλει θα επιτρέψουν καλύτερη διαχείριση και αποφυγή των, επι των επεισοδίων. Focus λοιπόν. Ο ορισμός των interface και ασφάλειες, ε, ασφαλιστικές δικλείδες. Βέβαια η φύση του προβλήματος είναι ακριβώς το ερώτημα. Μόνοι μας είμαστε. Όχι, αυτό δεν συμβαίνει. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αν δείτε τη στρατηγική που διαμορφώνουν οι ΙΠΑ, θα δείτε ότι η διαφορά εκεί μιλάνε για περισσότερο, μιλάνε περισσότερο για κυβερνοπόλεμο ή κυβερνοαδίκημα. Δεν, το, δεν είναι μια ορολογία που εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά πολλές από τις διαπιστώσεις είναι παρόμοιες και στις ΗΠΑ το βλέπουν από, πολλά, από πολλές οπτικές γωνίες. Σε πολλά κράτη-μέλη θα δείτε ότι μια συνεργασία μεταξύ Υπουργείων ήδη έχει ξεκινήσει ή ξεκινά το ζητάμε μάλιστα και ζητάμε ενίσχυση, ούτω ώστε να υπάρχει κοινή κοινά επεισόδια. Και δεν μπορεί να λέτε κατά πόσον αυτή θα είναι... Όταν έχεις μια απειλή δεν ξέρεις, μπορείς να πεις εκ των προτέρων ότι αυτή θα είναι μόνο κυβέρνο απειλή ή όχι. Και αυτό το βλέπουμε σε κράτη-μέλη. Θα χρειαστεί λοιπόν να έχουμε κοινέ προσεγγίσεις, έστω και αν αυτό είναι δύσκολο με σαφή ορισμό των interface και με διασφαλίσεις. Τονίζω επίσης ότι η στρατηγική δεν έχει να κάνει μόνο με την υιοθέτηση ενός νομοθετικού μέσου αλλά και με τις δράσεις που μπορεί να λάβει ο κόσμος και μάλιστα Τέθηκε η ερώτηση, τι μπορεί να κάνει ο κόσμος μόνος του, υπάρχει ετοιμότητα, υπάρχει δυνατότητα αυτόνομης διαχείρισης ε, κινδύνων. Πρόσφατα τον Οκτώβριο οργανώσαμε ένα μήνα επίγνωσης κυβερνοεπιθέσεων. Το κάνουμε δηλαδή, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη επίγνωση στον ιδιωτικό τομέα. Η στρατηγική έχει ήδη περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις Τώρα, για να γυρίσουμε στην οδηγία. Στην οδηγία σαφώς αναφέρεται ότι και ο ιδιωτικός, όχι μόνο ο δημόσιος τομέας, περιλαμβάνει παράγοντες με μεγάλη ευθύνη. Όταν θέλουμε να διαμορφώσουμε προσεγγίσεις ανάλυσης κινδύνου και προσεγγίσεις καταμερισμού των πληροφοριών, αλλά και με θέματα ε, προστασίας δεδομένων back-to-back, κάτι που δεν είναι πολύ μεγάλο βάρος και σίγουρα θα περιλαμβάνει και διαστάσεις αστικής ευθύνης αλλά και προστασία ε, βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλες αυτές οι διαστάσεις θα πρέπει να υπαχθούν στην ίδια οδηγία, αυτό είναι θέμα συζήτηση. Στην Αμερική βάλανε για παράδειγμα στην οδηγία ε, τις χημικές βιομηχανίες, αλλά δεν έβαλαν ε, τους Παρόχου ίντερνετ. εμεί του βάλαμε. Θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί υποχρεώσει, να υπάρχουν ειδικέ υποχρεώσει αυτών που παρέχουν software. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει να έχουν προδιαγραφέ για να παρέχουν λύσει στην αγορά με επαρκέ επίπεδο ποιότητα. Άρα, εξού και η ανάγκη συνεργασία με την ιδιωτική τομέα. Προφανώ δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα και άρα θα χρειαστούμε έρευνα και ανάπτυξη και παρεκκλίνω λίγο τις ομιλίες μου, υποστηρίζω αυτό που είπε λίγο ο Στίβ για την ασφάλεια και τον ιδιωτικό χώρο. Μήπως υπάρχει μια πρόκληση να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή η ισορροπία ασφάλειας και ιδιωτικής ζωής είναι ίδια, θα πρέπει να παραμείνει ίδια όπως είναι σήμερα ή να αλλάξει. Τονίζω πάντως ότι η οδηγία και η στρατηγική περιλαμβάνει ρητά μνήμα στην ε, προστασία των δεδομένων. Και η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη είχε εμπλακεί σημαντικά σε αυτό. Να τελειώσω. Γιατί tempus fugit. Πόροι Προφανώς μπορεί να βρεις πόρους από πολλούς τομείς. Και ευρωπαϊκή πόροι και ο ιδιωτικός τομέας. Η δουλειά δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει συνεισφορά, σημαντική συνεισφορά από τον ιδιωτικό τομέα. Βλέπουμε τον, την Ευρώπη 2020, μεγάλο εργαλείο, την, ε, το Connecting Europe, που παρέχουν διασυνοριακές ε, μορφές Τώρα, επαρκή πόροι υπάρχουν. Δύσκολο είναι για μας να πούμε πόσοι πόροι διατίθενται, γιατί πολλά γίνονται και σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βρούμε τη συνολοποίηση και του εθνικού επίπεδου. Η ερώτηση κρίσιμη είναι, έχουμε και προσωπικό με προσόντα, προσόντα όχι μόνο πανεπιστημιακού χαρακτήρα, αλλά και σε ενδιάμεσα επίπεδα. Κάποιον που μπορεί να δημιουργήσει ασφαλείς λύσεις, οδηγίες κατάρτισης και από τις εκθέσεις που διαβάσαμε σήμερα, διαπιστώνεται ότι θα υπάρξει μία μάχη για την ε, άντληση των σπάνιων πόρων ε, σε προσόντα που υπάρχουν στην αγορά. Και ξέρετε, στο παρελθόν, πριν από 10 χρόνια, δεν είχαμε επαρκή, επαρκή αριθμό ειδικών, γιατί κανείς δεν έκανε, κανένας δεν έκανε κυβερνοασφάλεια στο πανεπιστήμιο, δεν ήταν ενδιαφέρον. Τώρα άλλαξε η κατάσταση προς το αντίστροφο. Η απάντηση όμως που μπορώ να σας δώσω είναι ότι δεν έχουμε ακόμα επαρκή σπόρους στην Ευρώπη. Αυτά. Ευχαριστώ και τους τρεις σας για τις παρουσιάσεις σας. Είναι πρακτική της Επιτροπής Λίμπε να κάνουμε ακροάσεις και παρουσιάσεις. Διερμηνεύω και τα, συναισθήματα των μελών μας που ήταν σε αυτήν την συνεδρία και παρακολουθήσαν την παρουσίαση και τη συζήτηση που επακολούθησε. Είναι σαφές ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις σας λόγω του εξονυχιστικού και σε βάθος τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίσετε τα θέματα που διε... διελάβατε και λόγω και της ε, προσήλωσης που δείξατε στο πιο σημαντικό θέμα και το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και είμαστε σίγουροι ότι το θέμα αυτό θα βρίσκεται ψηλά στην ε, ατζέντα όλου του Κοινοβούλιου και όχι μοναχά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ευχάριστη η παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και κλείσαμε γέρος, γιατί τώρα έχουμε το επόμενο σημείο που είναι ακριβώς η παρουσίαση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στα σύννεφα. Στο σύννεφο, συγγνώμη, στο υπολογιστικό σύννεφος. Όπως έλεγα, τώρα περνάμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει να κάνει με την προστασία του ιδιωτικού βίου στο νέφος, το υπολογιστικό νέφος, το computer clouding. Και έχουμε την παρουσίαση μιας μελέτης από τον κύριο Μπάουτεν και τον καθηγητή Τιτιερ Πίγο, που καλωσορίζω εδώ. Ελάτε παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Εδώ θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση μετά την παρουσίαση της μελέτης που εκπώνησαν οι δύο ο κύριος Κάσφαν Πάουτερ και ο καθηγητής Τίτερ. Δικηγόρος. Όχι δικηγόρος. Θα μας παρουσιάσουν λοιπόν τα βρήματα της μελέτης αυτής και θα μας αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε. Προτείνω 20 λεπτά ο καθένας για να μας παρουσιάσετε τα αποτελέσματα και μετά θα δώσουμε το λόγο σε ευρωβουλευτές εδώ. «45 λεπτά θα διαθέσουμε, γιατί μετά έχουμε την εισηγήτρια την κυρία Σαρτζεντίνη και μετά θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Λοιπόν, ο καθηγητής Μπίγκο έχει πρώτο το λόγο. Έχουμε ετοιμάσει αυτές τις διαφάνειες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τίτλος είναι «Καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και προστασία του ιδιωτικού βίου στο υπολογιστικό νέφος». Είναι μια προπτική με πολλές διαστάσεις. Είμαστε μια ομάδα η οποία αποτελείται από διάφορους εμπειρογνώμονες, ε, δικηγόρους, αλλά και ειδικού ε, στις τεχνολογίες πληροφοριών. Είναι βέβαια τεχνικό το θέμα, αλλά όχι επειδή είναι τεχνικό πρέπει να είναι και δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Το θέμα αυτό δεν πρέπει να το χειρίζονται μόνο εμπειρογνώμονες και ειδικοί. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα από ό,τι δείχνουν. Τι είναι λοιπόν σημαντικό, και αυτό προσπαθώ να σας παρουσιάσω εδώ με τη δεύτερη διαφάνειά μου, Προσπαθώ λοιπόν να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Πρώτον, το θέμα είναι έχουμε περισσότερο έγκλημα. Δεύτερον, ε, χάνει κανείς τον έλεγχο των δεδομένων του. Τρίτον, οι νομικές πτυχές όσον αφορά το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων και ιδιαίτερα η αντίφαση μεταξύ των τάσεων ε, που υπάρχουν αν το κράτος λέει, θα δώσει προτεραιότητα στα δεδομένα στον πολίτη. Έπειτα υπάρχει το θέμα της δικαιοδοσίας και της ευθύνης και τέλος υπάρχει ρύθμιση της μεταβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες. Ας δούμε το θέμα λοιπόν του κυβερνοεγκλήματος και των ορίων του. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το cloud computing όσον αφορά το κυβερνοέγκλημα δεν εκτιμάει επαρκώς τα όρια του κυβερνοεγκλήματος όλα τα βάζουμε στο ίδιο καλάθι. Και αυτό είναι ο κίνδυνος, γιατί μπορείτε έτσι να έχετε σαφή όρια μεταξύ στοιχείων τα οποία είναι εντελώ διακριτά καταρχήν μεταξύ του. Υπάρχει το θέμα των πληροφοριών, υπάρχει το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών, το θέμα της αντιγκληματικής πολιτικής, το θέμα των απατών, τράπεζες κλπ. Είναι διαφορετικοί κόσμοι. Αν τους αναμίξετε μεταξύ τους, δημιουργείται πρόβλημα. Υπάρχει το κυβερνοέγκλημα, η κυβερνοαπάτη, υπάρχει όμως και η κυβερνοάμυνα, υπάρχουν ε, οι αγορές, υπάρχει το σαμποτάζ στον κυβερνοχώρο και διάφορες παράνομες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι πώς θα ανταλάβουμε υπόψη μας όλα αυτά γράφοντας ένα κείμενο. Δεν μπορεί, αν είσαι δικηγόρος, να τα λάβεις όλα υπόψη σου. Όταν τα μπερδεύει και έχεις και διαφορετικές πηγές, δεν μπορεί να έχεις καλό αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι είναι περίπλοκο να δουλέψεις λέγοντας ότι επειδή πρόκειται για τον χώρο, όλα τα βάζουμε μαζί. Το άλλο στοιχείο είναι η ιδιαιτερότητα του cloud computing σε σχέση με τον κυβερνοχώρο. Αυτή την ιδιαιτερότητα τη λαμβάνουμε υπόψη μας. Τα ευρωπαϊκά κείμενα δεν κάνουν την διάκριση αυτή γιατί αναφέρονται σε παραδοσιακές απειλές όταν μιλάνε για το νέφος. Ενώ όπως θα δούμε και αργότερα, πρόκειται για κάτι διαφορετικό και άρα θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Έπειτα υπάρχουν, ε, υπάρχει το ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος του, της ε, ΕΝΙΣΑ και της Europol όσον αφορά το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Η αποστολή και οι ορισμοί πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Το να μπερδεύουμε τα στοιχεία δεν μας οδηγούν σε έναν καλό ορισμό. Αντίθετα, δημιουργούνται επικαλύψεις και αποφεύγουμε τα προβλήματα. Αν δεν έχετε ξεκάθαρο ορισμό και ξεκάθαρες ευθύνες, τότε αντί να... τότε δεν δημιουργείται καλή συνεργασία, αλλά εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Κυβέρναγκλημα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι ο φόβος και το άλλο είναι το κόστος. Ο όρος κυβερνοέγκλημα έχει να κάνει με διάφορες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στην προηγούμενη παρουσίαση. Εγώ θέλω απλώ εδώ να καταδείξω ότι φυσικά το κυβερνοέγκλημα κατά είναι μπερδεμένο και έχει πολλές διαστάσεις, αλλά εξαρτάται από τις δραστηριότητες με τις οποίες εμείς ασχολούμεθα όταν μιλάμε για το κυβέρνο έγκλημα. Για τον Ευρωπαίο πολίτη, μπορούμε να μιλήσουμε για τις απάτες που γίνονται σε βάρος του. Έχουν γίνει υπολογισμοί 10 πένες το χρόνο κατά κεφαλή. Αν όμως θέλετε να το αποφύγετε μέσω μεθόδων ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, τότε θα ξοδέψετε 60 ε, λίρες, λίρες όχι, 60 λίρες θα ξοδέψετε τότε. Ο φόβος είναι θεμητός, έχει όντως βάση ή πρόκειται για το φόβο των ε, πολιτικών. Όσον αφορά γενικά το κυβέρνο έγκλημα. Όντως κάποια στοιχεία του είναι πράγματι σημαντικά, κάποια άλλα όμως είναι λιγότερο σημαντικά. Που θα ήταν προτιμότερο να αντιμετωπιστούν με την ε, καταστολή και όχι με την πρόληψη. Τι τώρα δεν βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης. Είναι την ε, πρόκληση που έχει να κάνει με τον ιδιωτικό βίο. Το cloud computing ιδιαίτερα το υποτιμάμε. Και αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που διαπιστώνουμε όταν γίνονται συζητήσεις μεταξύ ειδικών. Το μοντέλο που έχουμε των τελευταίων 40 χρόνων για τη μεταβίβαση δεδομένων είναι τελείως διαφορετικό από τη σημερινή κατάσταση. Ποιος είναι ο κίνδυνος για τον καταναλωτή είναι ότι το clouding μπορεί να μην χρησιμοποιεί σωστά τα δεδομένα τα οποία βρίσκονται στα κέντρα του. Οπότε για τα δικαιώματα των καταναλωτών προφανώς υπάρχει το πρόβλημα του ποιος ιδιωτικός φορέας τελικά χειρίζεται τα δεδομένα του. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα του ατόμου και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να προστατεύει τα δομένα. Το οποιοδήποτε σχετικό παράπτωμα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Γιατί όμως δεν συμβαίνει αυτό, δεν είναι προτεραιότητα. Γιατί για άλλη μια φορά φαίνεται ότι πρέπει κανείς να διαλέξει πού θα επικεντρωθεί στην κυβερνοασφάλεια, όπου εκεί τίθεται το θέμα της εθνικής ασφάλειας, άμυνα, έγκλημα, αστυνομία, εκεί θα επικεντρωθούμε ή θα επικεντρωθούμε στον πολίτη έχετε δύο απόψεις αντίθετες μεταξύ τους όταν αναλύει κανείς τη σχέση των ε, επιχειρήσεων Το στοιχείο κλειδί εδώ είναι ότι οι περισσότερες υπηρεσίες θέλουν μια σφαιρική ρύθμιση του διαδικτύου. γιατί έτσι μπορείτε να έχετε κοινέ στρατηγικέ, οι οποίες να μην είναι μόνο εθνικές ή ευρωπαϊκές, αλλά να ισχύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό ακριβώ είναι που βρίσκεται και στην καρδιά της συζήτηση. Αν κοιτάξετε στην επόμενη διαφάνεια εδώ τι γίνεται με το IP και το κυβέρνο έγκλημα σε σχέση με το computer clouding, απαιτούνται κανόνες οι οποίες να επιτρέπουν τη σύνδεση των ατόμων με τις διευθύνσεις των ε, παρόχων. Αυτό εν μέρη θα μπορούσε να λύσει κάποια προβλήματα, τουλάχιστον θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα να λυθούν κάποια προβλήματα. Τα πιο γενικά. Δημιουργεί όμως και πολλές δυσκολίες για την σχέση μεταξύ χωρών, επιχειρήσεων, συστημάτων. Εδώ είναι διαλειτουργικότητα. Και η δημιουργία πολλών και διαφορετικών συστημάτων σε διαφορετικά μέρη. Αυτό λοιπόν πρέπει να αποτελέσει ένα κομμάτι της συζήτησης. Και γιατί Έχουμε το θέμα της διάθεσης δεδομένων και της προστασίας των δεδομένων στο cloud computing. Και είναι πολύ περίεργο που η ορολογία των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, ακριβώς είναι στο κέντρο της συζήτησης αυτής. Έχει να κάνει με τις χώρες, με την ασφάλεια των χωρών, των επιχειρήσεων κλπ. Το άτομο όμως πού βρίσκεται, δεν βρίσκεται πουθενά. Και αυτό εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το άτομο να δούμε. Το άτομο ως άτομο και όχι ως καταναλωτή. Το άτομο ως πολίτη. Αυτό το στοιχείο κλειδί είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Δεν το αντιμετωπίζουμε όμως, γιατί επικεντρωνόμαστε στην εθνική ασφάλεια, στο έγκλημα και όχι στο άτομο. Και άρα βερδεύουμε τις προτεραιότητές μας. Λέμε ότι η προτεραιότητα θα είναι ή ένα ή το άλλο. Αν δούμε την προστασία των πολιτών από το έγκλημα ή από την κατάχρηση των δεδομένων του από κάποια όργανα, από κάποιες επιχειρήσεις, αυτό είναι κάτι τελούς διαφορετικό. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε εξετάσει επαρκώς. Και θα τελειώσω με την προστασία δεδομένων με το εξής η πρόκληση αυτή της προστασίας των δεδομένων, πώς θα την αντιμετωπίσουμε, πώς θα την αντιμετωπίσει το computer clouding και ποιος θα προστατεύσει τα δεδομένα των πολιτών όταν αυτά θα τυχαίνουν προστασίας βάσει νομοθεσίας τρίτων χωρών. Ο συνάδελφος όμως θα επεκταθεί περισσότερο. Ευχαριστούμε καθηγητά Μπίγκοφ, κύριε Μπάρτνερ, η σειρά σας. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Μπίγκοφ γιατί έθεσε τα διακλαδικά ζητήματα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω τώρα είναι να εστιάσω σε μια συγκεκριμένη πτυχή της έκθεσής μας με πιο συγκεκριμένους όρους. Μπορεί να σας βοηθήσει να σκεφτούμε τους κλάδους που μας έχουν απασχολήσει. Μιλήσαμε για το κυβερνοέγκλημα, αλλά δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε το πακέτο για, το, για την κυβερνοασφάλεια σε επίπεδο ερωτήσεων φυσικά θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εδώ. Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει, όπως είπε ο καθηγητής Μπίγκοφ, θέματα εθνικής ασφάλειας που είναι λεπτά θέματα. Υπάρχει και ένας τρίτος χώρος που είναι της συλλογής πληροφοριών, ευαισθήτων πληροφοριών από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να γυρίσουμε προς τα πίσω και να καταλάβουμε ότι τα θέματα εθνικής ασφάλειας είναι εθνικά θέματα, αυτό είναι και μέσα στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι πολύ θεμητό για αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ενέργειες συλλογής πληροφοριών τρίτων χωρών που είναι παράνομες βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. αν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην προηγούμενη διαφάνεια, η εικόνα αυτή είναι μια εικόνα νέφους ενός κέντρου δεδομένων και στα δεξιά βλέπετε μια αίθουσα η οποία έχει δημιουργηθεί σε ένα κέντρο ε, τηλεπικοινωνιακής ε, τηλεπικοινωνία στο Σαν Φρανσίσκο και το ερώτημα είναι αν υπάρχει μια αίθουσα σαν τη δεξιά σε ένα κέντρο δεδομένων όπως υπάρχει και η αριστερή αίθουσα. Όταν μιλάμε λοιπόν για, την, για το υπολογιστικό νέφος, σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ένας χώρος να αποθηκεύουμε τα email μας και τις φωτογραφίες. Αλλά η ατζέντα για τους επιχειρηματίες και τις κυβερνήσεις είναι πιο σημαντική. Γιατί μέχρι πρόσφατα, αν μια κυβέρνηση, μια επιχείρηση <clears throat> θέλαν να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών, θα το κάνανε χρησιμοποιώντας λογισμικό και υλικό που βρίσκεται μέσα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αλλά το πρόβλημα που προκύπτει από τη βιομηχανική κρίση του υπολογιστικού νέφους είναι η δυνητική μετακίνηση όλων των ευρωπαϊκών στοιχείων στο νέφος, όχι για αποθήκευση αλλά για επεξεργασία γιατί το πλεονέκτημα του νέφους για επεξεργασία είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ικανότητα υπολογισμού <clears throat> χιλιάδων υπολογιστών για να μπορεί κανείς να εργάζεται εν παραλίλω πάνω στα ίδια στοιχεία και αυτό είναι πιο μεγάλο πλεονέκτημα του νέφους από την ικανότητα αποθήκευσης. Επόμενη διαφάνεια. Πρέπει να αναφερθώ σε μία χώρα δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα αυτά τα θέματα χωρίς να μιλήσω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει τη μεγαλύτερη βιομηχανική ικανότητα και σε software και σε hardware, λογισμικό και υλικό για το υπολογιστικό νέφος. Το 2003 ένας τεχνικός στην AT&T στο Σαν Φρανσίσκο ανακάλυψε ότι υπήρχε μια μυστική αίθουσα στο κέντρο ε, διακομισμού που ουσιαστικά περνούσε από εκεί ο, η ροή δεδομένων της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών και η παροχετευμένη αυτή ροή εξεταζόταν από ένα ειδικό σύστημα <clears throat> και ένα τμήμα από αυτό μετά από ανάλυση περνούσε στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η ιστορία έγινε γνωστή μόνο το 2005, δημοσιεύτηκε στους New York Times και μετά υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι έκρουσαν τον κόνδωνα του κινδύνου και από την FBI και από την ε, NSA, την ε, Υπηρεσία Έθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, που τόνισαν όλοι αυτοί ότι ήταν παρακολούθηση των ίδιων των πολιτών των ΗΠΑ με παράνομο τρόπο το 2007. Με την, ε, μετά από την διαμάχη που ακολούθησε, όλες αυτές οι δραστηριότητες έγιναν νόμιμες με, το λεγόμενο νόμο «Προστατεύστε την Αμερική» που ουσιαστικά νομιμοποίησε ένα νέο παράδειγμα συλλογής δεδομένων, δηλαδή το ότι μπορεί να συλλέγονται όλα τα δεδομένα και να αναλύονται στη συνέχεια. Επίσης, ο νόμος αυτός στις ΗΠΑ ε, περιέχει ειδικές προστασίες για τους πολίτες των ΗΠΑ. Όλη η διαμάχη αφορούσε τελικά το, τα δικαιώματα των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν έλεγε τίποτα για τα δικαιώματα ξένων πολιτών. Αν μπορώ να περάσω στην επόμενη διαφάνεια τώρα, το 2008, πριν εκλεγεί ο πρόεδρος Ομπάμα και τα δύο κόμματα στη, στο Αμερικανικό Κογκρέσο αντιμετωπίσαν τα θέματα αυτά με την τροπολογία ΦΙΖΑ του 2008 που τροποποιεί νομοθεσία του 1978. Και το τμήμα της το 1881α προβλέπει την συλλογή δεδομένων από ξένες πηγές αντιμετωπίζει μονάχα του, τον υπόλοιπο κόσμο μη Αμερικανούς πολίτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει μια συνολική έγκριση για μέχρι ένα χρόνο, ζητά ε, να υπάρξει ελαχιστοποίηση στοιχείων για πολίτες Ηνωμένων Πολιτών μετά τη συλλογή δεδομένων και λέει ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν απόλυτα μυστικά με διάφορες ε, ποινές εάν δεν τηρηθεί το εμπιστευτικό και λέει ότι αυτά πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο ο οποίος συνάδει με την τέταρτη ε, τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος που προστατεύει την ιδιωτική ζωή. Τι είναι όμως τώρα αυτή η συλλογή ε, πληροφοριών, ευαισθητών πληροφοριών από ξένους χώρους. Αντιμετωπίζει θέματα σαμποτάζ, τρομοκρατία, σοβαρού εγκλήματος όπως θα περίμενε κανείς, αλλά περιλαμβάνει και πληροφορίες σε σχέση με πολιτικές οργανώσεις εκτός των ΗΠΑ ή απλώς για ξένα εδάφη που μπορούν να έχουν σχέση με την ε, άσκηση της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ευρύτατος λοιπόν αυτός ο ορισμός. Και αν συγκρίνεται αυτή την νομοθεσία με την νομοθεσία για την εθνική ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών δεν βλέπει κανείς πουθενά μια τόσο ευρεία εντολή για πολιτική παρακολούθηση το τμήμα 1881α της Φάιζα συνδυάζει για πρώτη φορά τρία στοιχεία που μέχρι τώρα ήταν σε διαφορετικά ε, νομοθετήματα. Για πρώτη φορά συνενώνται το 2008 πρώτον το ότι στοχοποιούνται οι, πολίτες, οι μη πολίτες των ΗΠΑ, ο υπόλοιπο κόσμος δηλαδή. Δεύτερον, αφορά τις λεγόμενες εξαποστάσεως υπηρεσίες υπολογισμού, και αυτό είναι καινούριο. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζει, εφαρμόζεται στο υπολογιστικό νέφος. Δεν πρόκειται μονάχα για εταιρείε τηλεπικοινωνιών όπως η AT&T. Σημαίνει ότι μεγάλη ε, παροχή όπως η Microsoft ή η Google μπορούν, πρέπει, μπορούν να, ζη, να τους ζητηθεί να συμμορφωθούν με αυτήν την νομοθεσία. Αν χρησιμοποιείτε παραγωγή χάρη κρυπτογράφηση για να προστατευτούν τα στοιχεία σας από τον υπολογιστή σας στο νέφος, δεν υπάρχει καμία προστασία γιατί οι Αμερικανικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κέντρο αυτό ε, δεδομένων και να έχουν πρόσβαση για τα στοιχεία σας. Αλλά αυτό, σας λέω και πάλι, το θέμα δεν είναι η αποθήκευση, αλλά η ικανότητα μαζικής υπολογιστικής επεξεργασίας. Και τρίτον, δεν έχουν να κάνουν τίποτα αυτά με εγκληματικότητα ή με την εθνική ασφάλεια μπορεί να υπάρξει αποκλειστικά και μόνο πολιτική παρακολούθηση για να υποστηριχθούν οι στόχοι εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Αναφέρθηκα στο 1881, υπήρχε η ρήτρα ότι αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι συμβατός με την τέταρτη τροπολογία και είδατε πολλές φορές στοιχεία από τις ε, υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας υπενθυμίζω ότι πουθενά δεν αναφέρεται το οτιδήποτε έλεγα ως τώρα. Μέχρι τώρα υπήρξε απόλυτη σιωπή ασυρμάτου από την πλευρά της, των Πολιτειών για όλα αυτά τα θέματα από την έκδοση της ΦΑΙΖΑ Και προέκυψε αποσπασματικά τα τελευταία χρόνια ότι η τέταρτη τροπολογία δεν προστατεύει παρά μόνο τους Αμερικανούς πολίτες. Δεν προστατεύει ανθρώπους που δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών που μπαίνουν στο υπολογιστικό νέφος μπορούν να υποβάλλονται σε παρακολούθηση για καθαρά πολιτικούς στόχους και μόνο. Δεν θα τα συζητήσω τα θέματα ιδιαίτερα λεπτομεριακά, αλλά αυτό που σας δείχνει αυτή η διαφάνεια είναι ότι αν δείτε τις τεχνικές βάσεις του νέφους του υπολογιστικού για παράλληλη επεξεργασία υπάρχει ένα κίνητο για τις κυβερνήσεις αυτές που θέλουν να κάνουν ε, συστηματική παρακολούθηση για τον έφος. Θα πρέπει να πάνε και να ζητήσουν από τη Microsoft και την Google να δημιουργήσουν μέσα στο λογισμικό τους την δυνατότητα παρακολούθησης. Θα πρέπει να αναπαραίτητο να υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσα στο ίδιο τον έφος. Δεν έχω το χρόνο να σας τα παρουσιάσω αυτά, αλλά θέλετε μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις. Και αυτή η διαφάνεια καταδεικνύει ότι δεν μιλάμε για μια αίτηση για δεδομένα. Δεν μιλάμε όπως πιστεύουν οι αρχές προστασίας δεδομένων ή όταν συζητήθηκε η, η νομοθεσία περί πατριωτικής προστασίας δεν είναι ένα νομικό εργαλείο για να ζητείτε αίτηση κάποιων δεδομένων. Αυτή είναι μια κατάσταση όπου υπάρχει μαζική παρακολούθηση η οποία γίνεται συγχρόνως και συνεχώς για όλες τις ροές δεδομένων. Και αυτό το γράφημα δείχνει ήδη από το 2006 από την Ένωση Αστικών Δικαιωμάτων τις ροές αυτές σε διάφορα κέντρα, γιατί δεν ήταν μόνο το κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, αλλά διάφορα κέντρα στις υποδομές των ΗΠΑ. Το επόμενο. Ίσως λοιπόν με ελαφρό τρόπο το έχω παρουσιάσει αυτό σαν μια γραμμή μαζινό στον κυβερνόχωρο. Τα μέλη του Κοινοβουλίου βέβαια έχουν ε, διαπραγματευτεί διαφυλάξεις για το PNR και το SWIFT. Αλλά από αυτά που σας είπα, όλες αυτές οι συμφωνίες μπορούν να παρακαμφθούν και να υπάρχει άμεση και μαζική παρακολούθηση όταν όλα αυτά τα στοιχεία μπαίνουν στο υπολογιστικό νέφος. πριν από 18 μήνε ακόμα δεν ξέραν οι αρμόδιες αρχέ για τα θέματα αυτά. του ενημέρωσα ιδιωτικά τον ε, Ιούνιο του 2012 το, η ομάδα εργασίας του ΑΦ 29 έδωσε μια γνωμοδότηση στο, για το υπολογιστικό νέφος. Μιλάνε για την πρόσβαση των εθνικών υπηρεσιών για την ε, εφαρμογή του νόμου και τόνισαν ότι, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν ε, συμφωνίες συνθήκες με άλλες χώρες για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η πρόσβαση σε δεδομένα. Η λύση όμως που προσφέρουν νομίζω ότι είναι ανοιχτή σε επικρίσεις. Δεν έχω και πάλι το χρόνο να σας πω γιατί γίνεται ακριβώς αυτό. Αλλά η νομική λύση που δίνουν δεν αποτελεί λύση. Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στο πακέτο για προστασία δεδομένων έχουμε τους λεγόμενους δεσμευτικούς Κανόνε για τι επιχειρήσει σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω αυτά, βρίσκονται στην εκθεσή μα πιο λεπτομερώς, αλλά είναι ένα νομικό μηχανισμό ο οποίο έχει δημιουργηθεί μεταξύ των αρχών προστασία δεδομένων και των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια για να νομιοποιήσει ροέ ε, προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών στο νέφο. Και όταν βλέπουμε τη διατύπωση του άρθρου 29 για όλα αυτά, επόμενη διαφάνεια, βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη και αρκόπορτες για όλα αυτά. Όταν δει κανείς τα ψηλά γράμματα του, τι είπε το άρθρο 29 για τις ε, προϋποθέσεις αυτές, προβλέπεται η εφαρμογή ε, νομοθεσίας όπως η πράξη για την προστασία της πατρίδας των ΗΠΑ ή η ΦΑΙΖΑ. Όλα αυτά δεν μπορούν να εμποδιστούν από το πακέτο για την ασφάλεια στον κυβερνόχρονο όπως έχει τώρα. Για όλα αυτά λοιπόν πιστεύουμε ότι όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις λεγόμενες συζητήσεις ε, συνολικές ε, στο πλαίσιο της εφαρμογής ε, του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βασική θέση των ΗΠΑ είναι ότι αυτή η συμφωνία, ομπρέλα όπως αποκαλείται, δεν θα περιλαμβάνει, δεν θα καλύπτει μεταφορές από ιδιώτη σε ιδιώτη που συμβαίνει με το cloud. Συνοπτικά, συνοψίζοντας μάλλον, η κατάσταση έχει ως εξής. Η παρακολούθηση του cloud είναι για όλη την Ένωση. Θυμάστε το Εσελον, αλλά το εσελόν αφορούσε μόνο επικοινωνία, ενώ εδώ μιλάει για παρακολούθηση όλων των δεδομένων της Ένωσης που μπαίνουν στο cloud. Όπως σας είπα, η κρυπτογράφηση δεν ε, έχει νόημα, διότι αποκρυπτογραφείται αυτόματα από τον πάροχο του cloud. Προφανώς αν θέλετε να κάνετε μόνο αποθήκευση μπορείτε να το, να το κρυπτογραφήσετε οι ίδιοι. Η παρακολούθηση από τρίτες χώρες ή τρίτες κυβερνήσεις είναι τελείως διαφορετικό θέμα από αυτές των ε, κυβερνήσεων της Ένωσης. Κυρίως γιατί δεν υπάρχει η τήρηση των ε, του χάρη των θεμελιών δικαιωμάτων. Άρα, από το 2008 είναι νόμιμη η παρακολούθηση των δεδομένων των πολιτών της Ένωσης και το χειρότερο είναι ότι κανείς δεν το έμαθε, δεν το, διαπίστωσε, δεν το έλαβε υπόψη του, κανείς δεν το πρόσεξε. Αυτό είναι σύλληπτο. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι στη διατύπωση του κανονισμού προστασίας δεδομένων τα παραθυράκια που το επιτρέπουν ήδη υπάρχουν από τις αρχές ε, προστασίας δεδομένων που υποτίθεται ότι μας προστατεύουν. Η έκθεσή μα έκανε, έδωσε μια... Τους πάντων έφερε την προσοχή του κοινού τις τελευταίες εβδομάδες. Αν δείτε τα Twitter και τα ρεπορτάζ των εφημερίδων. Η κοινή γνώμη ωστόσο στην Ευρώπη είναι ε, έχει μείνει αποσβολωμένη. Δεν μπορεί να καταλάβει πως ένας μηχανισμός προστασίας δεδομένων φτάνει σε μια κατάσταση όπου όχι μόνο αγνοεί, αλλά επιτρέπει η παρακολούθηση. Ζήτω συγγνώμη, νομίζω ότι μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή παρά αυτά. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο ομιλητές. Έχουμε και λίγα λεπτά και να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Κάποιος συνάδελφος θέλει να θέσει ερώτηση. Κύριε Σαρτζαντίνη και η κυρία Ιντβελτ. Ευχαριστώ. Για τη δεύτερη παρουσίαση θα κάνω σχόλιο. Η πρώτη ταυτιζόταν εμπολής με τις παρατηρήσεις που έκανα στην προγενέστερη παρέμβασή μου για την κυβερνοασφάλεια. Χαίρομαι πολύ που θέσατε το θέμα αυτό, γιατί όπως ξέρετε η πρώτη φορά που υπέβαλα μια κοινοβουλευτική ερώτηση το 2007 σχετικά, και νωρίτερα ίσως δεν θυμάμαι, και εγώ όπως και εσείς πραγματικά μένω ενεός που κανείς δεν το παρακολούθησε. Και δεν είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και αν δεν ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά άλλη χώρα που δεν χρειάζεται καν νομοθεσία για κάτι τέτοιο. Και μην ξεχνάτε ότι ε, όλο και οι περισσότερε επιχειρήσει εγκαθίστανται εκεί και όλο και οι περισσότερε χώρε θα ενδιαφέρονται. Θέλω να τονίσω ότι το θέμα εδώ δεν είναι τεχνικό. Το cloud απλά το επιδεινώνει. Το βασικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα δικαιοδοσίας και αρχεία σε χαρτί να ήταν, το ίδιο πρόβλημα θα ήταν. Μια τρίτη χώρα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρεί ότι τα στοιχεία και τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ευρωπαϊκό έδαφος υπάγονται στη δική του δικαιοδοσία γιατί αυτοί έχουν δικό του ορισμό της δικαιοδοσίας. Μπορεί να γκρινιάζουμε για τη Ρωσία, την Αμερική, την Κίνα αλλά το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Εμείς το είπαμε και το ξανάπαμε χιλιάδες φορές στην Επιτροπή. Με ερωτήσεις από το 2007 σας είπα και πριν από αυτό. Η Επιτροπή μέχρι τώρα δεν έχει πει τίποτα. κλείνει τα μάτια της. Είτε γιατί φοβούνται να συγκρουστούν με τους Αμερικάνους ή δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν. Η Επιτροπή λέει ότι το πρόβλημα θα λυθεί με το νέο κανονισμό. Όχι δεν θα λύθει το πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις δεν προστατεύουν, δεν προσπίζουν τα συμφέροντα των πολιτών. Ε, ο, νόμος, ο πατριωτικός νόμος, και το είχαμε πει και στην κυβέρνηση της Ολλανδίας και αλλού τέθηκε ενδεχομένως, δεν ξέρω. Λόγω του πατριωτικού νόμου, τμήμα του είναι το Βάιζα, η εταιρεία που ετοιμάζει Ολλανδικά διαβατήρια που περιλαμβάνει δακτυλικά αποτυπώματα των δανών πολιτών τα στοιχεία αυτό είναι προσπελάσιμα στις αρχές των ΗΠΑ. Τώρα δημιουργούμε ένα σύστημα ιατρικών δεδομένων που θα το διαχειρίζεται μια εταιρεία που δεν μας εκπλήσει έχει και παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα και αυτή υπάγεται στις διατάξεις του πατριωτικού νόμου. Χαίρο που πήρε δημοσιότητα η έκθεσή σας, γιατί ελπίζω κάποιος στην Επιτροπή να λάβει σοβαρά το θέμα υπόψη και να δώσει απάντηση. Πρέπει να δώσει απάντηση, δεν μπορούν να σιωπούν τώρα που τους δώσετε τόσο υλικό και τους υποχρεώνετε τώρα να απαντήσουν. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Θα επανέλθω για το cloud computing ε, μετά. Κύριε Μπάουρεν, είπατε και το έχετε ξαναπεί σας, είχα ακούσει παλιότερα, ότι η οδηγία για την προστασία των δεδομένων δεν καλύπτει τα κενά που πρέπει να καλυφθούν για να εξασφαλιστούν τα δεδομένα μας. Μπορεί να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος γιατί ο Σονούπο τελειώνει η λίγη προθεσμία για την υποβολή των υπολογιών. Η κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ όπως και οι συνάδελφοι έχω μείνει έκθαμβη από τις εξηγήσει που είδαμε. Όποτε μιλούσαμε για το cloud, αυτό φαινόταν ένα ταμπού. Κανείς δεν ξέρει τι είναι, που βρίσκεται, τι, τι περιλαμβάνει. Είναι απλό το θέμα. Μετά τις εξηγήσει που είχαμε σήμερα, δεν φαίνεται ότι στην Ευρώπη υπήρχε ενδιαφέρον να μπει πιο διεξοδικά η μελέτη στο θέμα αυτό. Ίσως είναι σφαλμένη η προσέγγιση. Όλο το απόγευμα μιλούσαμε για, κυβερνο, για το κυβερνοέγκλημα. Δεν μιλάμε όμως για τα δικαιώματα των πολιτών που οι πολίτες είναι αυτοί που δίνουν τα στοιχεία τους χωρίς να συνενούν. Αυτό είναι πιο συγκεκριμένο βαθύ πρόβλημα. Δεν είναι εγκληματικότητα οι εγκληματίες μπορεί να χρησιμοποιήσουν προφανώς την τεχνολογία αυτή. Αλλά εμείς μιλάμε για κάτι πιο θεμελιακό όπως είπατε. Και αυτό το το βλέπει η Κομισιόν και το αγνοεί. Μιλάμε για προστασία δεδομένων, για ολόκληρο πακέτο προστασίας δεδομένων, χωρί να μιλάμε για το cloud. δίνουμε τα αρχεία μας σε μια χώρα που δεν ξέρουμε καν ποια είναι γιατί ε, που ξέρουμε που θα είναι φυσικά αυτές οι βάσεις δεδομένων. Ξέρουμε τώρα σήμερα, μετά από αυτό που μας είπατε, ξέρουμε τι μπορεί να είναι στις Ηνωμένες Το θέμα αυτό δεν πρέπει να το δούμε. Είναι θέμα διεθνούς δικαίου. Πρέπει να το αντιμετωπίσει η Επιτροπή είτε με αμοιβαία συνεργασία, αλλά ε, σε κάποια φάση στο πλαίσιο της προστασίας δεδομένων πρέπει να μιλάμε για το cloud computing. Τι είναι αυτό που επήγει περισσότερο να κάνουμε στο θέμα αυτό του cloud. Γιατί μιλάμε για ε, ευθύνες. Ο ένας είναι υπεύθυνος, ο άλλος είναι αρμόδιος ε, και κανείς δεν κάνει τίποτα. Δίνουμε σε τρίτες χώρες χωρίς έλεγχο τα στοιχεία. Είναι δυνατόν να διπάρξουν κάποια σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα για να μπορέσουμε να λάβουμε, να, προστατεύσουμε τη διάσταση που αυτή και πραγματικά αυτό είναι εξαιρετικά επιούν και σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσετε. Απαντήσεις. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να θέλει το λόγο. Ο κύριος, ο καθηγητής Μπίγκο ή ο κύριος Μπάουντεν. Πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτον, να συγχαρώ την κυρία Τεβέλτ για τη δουλειά της στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι από ό,τι ξέρω δούλεψε για το θέμα αυτό περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον ε, ευρωβουλευτή. Αυτό που σας μιλάω, αυτό για το οποίο σας μίλησε εδώ το Φάιζα, είναι άσχετο με τον, το Patriot Act. Η έκθεση αυτό που θέλει να πει είναι ότι ο νόμος για την τροποποίηση, ο Φάιζα Amendment Act, ε, το, ε, ε, είναι ξεχωριστός νόμος και αν δεν είσαι Αμερικανός πολίτης είναι ακόμα χειρότερος Τώρα, για τις προθεσμίες ε, που αναφέρατε, στη σελίδα 48 της έκθεσης κάνουμε κάποιες ε, προκατακτικές συστάσεις και θα σας τις συνοψίσω. Πρώτον, να μην εφαρμόζουμε τις παρεκκλήσεις για την ε, μεταφορά αρμοδιοτήτων εκτός ένωσης για το cloud. Άρα δεν είναι μόνο θέμα δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, είναι θέματα συμβάσεων, όποια μεταφορά γίνεται με την υφιστάμενη παρέκκληση δεν προστατεύει πολιτική ε, παρακολούθηση μέσω του Βάισε και αυτό το ξέρουν οι αρχές προστασίας δεδομένων. Πολλές από τις αρχές δεν ήταν ε, ευχαριστημένες με την έννοια του ασφαλούς ε, καταφυγίου, του safe harbor, αλλά υποχρεώθηκαν το την να το εφαρμόσουν. Υπογραμμίζω ότι η εφαρμογή του VISA στο cloud computing είναι που δημιουργεί ανησυχία. Μια άλλη σύσταση που κάνουμε είναι ότι απαιτούνται πιο γρήγορες και άμεσες μελέτες ε, έρευνες ε, επιστημονικές γιατί πολύ λίγοι επιστήμονες και πανεπιστημιακοί έκαναν ε, έρευνα συγκριτικής νομοθεσίας, όχι μόνο με τη ΣΥΠΑ αλλά και με άλλες χώρες. Δεν υπάρχει συγκριτική ανάλυση, ούτε καν πλήρης ανάλυση των ΗΠΑ. Υπάρχουν, η, η δική του τομέα είναι δύο-τρεις και σχεδόν κατά Σα τα είπα αυτά που σα τα είπα σήμερα, γιατί η αρχική πρόταση που είχε γίνει για την ημερήσια διάταξη δεν περιέλαβε κάτι τέτοιο. Αν μη τι άλλο θα έπρεπε να προειδοποιηθούν οι πολίτες της Ένωσης ότι όταν περνούν δεδομένα τους στο cloud που μπορεί να υπαχθεί σε δικαιοδοσία ενός άλλου κράτους ενδέχεται οι πολιτικές θέσεις του, για παράδειγμα να ε, γίνουν γνωστές στις αρχές της χώρας αυτής. περιέργως μία από τις ε, πιο ικανές δομές προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη είναι η περιφερειακή δομή δεδομένων του Σλέσβικ Χολστάιντ που ήταν η μόνη που έκανε μία τέτοια ενημέρωση στους πολίτες της του Σλέσβικ Χολστάιντ. Τελευταία σύσταση. Όπως είπε και η κυρία Νίτενβέλ, δυστυχώς δεν υπάρχει νομική προστασία ή τεχνική προσταγγίηση ότι μπορεί τα στοιχεία σου να χρησιμοποιηθούν και να γίνει αυτό που είδατε στο κέντρο της AT&T. Μπορεί να γίνει και δεν μπορείς να προστατευτείς. Δεν υπάρχει έλεγκτης που, κάνει, που, που, που, που συμπληρώνει τετραγωνάκια ναι, ναι, ναι. Κανείς δεν θα σου πει ότι κάτι τέτοιο έγινε. Η μόνη εναλλακτική λύση είναι να υπάρξει μία ογκώδης δομή αποθήκευσης cloud στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε όχι μόνο το hardware αλλά και το software και κατά την άποψή μου πρέπει να είναι open source software, ανοιχτό. Και προτείναμε ένα στόχο 5% του δημοσίου να, γι, να πηγαίνει στο cloud μέχρι το 2020. Αυτό ευθυγραμμίζεται και με άλλους στόχους ε, που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πληροφορική στο παρελθόν. Θα επανέλθω δυστυχώ, ωστόσο, στη βασική παρατήρηση. Με εκπλήσει το ότι το ζήτημα αυτό έχει αγνοηθεί σημαντικά και από την Επιτροπή και από τις αρχές προστασίας δεδομένων. Ευχαριστούμε. Ο καθηγητής Μπίγκο. Κάτι ακόμα. πρέπει να είμαστε σαφείς για το εξής, ότι ένας Ευρωπαίος πολίτης ε, δεν έχει καμία επιλογή αν μια εταιρεία βγάζει τα προσωπικά του στοιχεία στο υπολογιστικό νέφος. Οι πολίτες λοιπόν δεν έχουν τη δυνατότητα να ξέρουν αν μια εταιρεία το κάνει αυτό για δικούς τους λόγους. Γιατί και αυτοί δεν κατανοούν ποιο είναι το πρόβλημα που αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις εταιρείε. Ευχαριστώ, Λέω ο Πρόεδρος. Ήταν σαφές αυτό. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το οποίο και αυτό αφορά τα θέματα του πακέτου για την κυβέρνο ασφάλεια. Περνάμε στο σημείο 14 για τις δυνατότητες του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη. Η κυρία Σαρτζεντίνη είναι η αρμόδια. Καταρχήν όμως θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους δύο μιλητές μας για σήμερα το απόγευμα για την παρουσία, τον κύριο Μπίκο και τον κύριο Μπάουντεν. Κυρία Σαρτζεντίνη, τώρα είναι η σειρά σας. Να παρουσιάσετε το την ε, γνωμοδότησή σας για την επόμενη μισή ώρα. Δεν θα μιλήσω για μισή ώρα. Δεν περιμένετε μισή ώρα να μιλήσω. Όχι, όχι. Το σημείο σας μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα μετά, μην νομίζετε. Έχετε το λόγο, κύριε Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Μπίγκορ. Βλέπω ότι είναι ακόμα εδώ και παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν από λίγο ήρθε κάποιος από την Amazon ε, Ευρώπη σε μένα και εγώ νόμιζα ότι πουλούσαν βιβλία και DVDs και ναι μεν πουλούν βιβλία και DVDs, αλλά και χώρο στο νέφος. Αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους. Και εγώ ρώτησα, αν εγώ νοικιάσω χώρο στο νέφος σας, ήμουν αφελής βλέπετε ακόμα, ε, έτσι ένα νέφος πάνω από την Ευρώπη σκεφτόμουν, θα είμαι ασφαλή. Ναι, ναι, μπορούμε να σα το εξασφαλίσουμε. Όντω, πρόκειται για ένα έφο πάνω από την Ευρώπη, οπότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα με τα δεδομένα σα. Όταν έφυγε όμω η κυρία αυτή, κατάλαβα ότι δεν με βοηθάει καθόλου, γιατί η Amazon είναι αμερικανική επιχείρηση. Ετοιμάζω γνωμοδότηση λοιπόν Γνωμοδοτούμε προς την ε, Ήτρε. υπάρχει το άρθρο 50, υπάρχει το θέμα της προστασίας των δεδομένων και το θέμα του κυβερνοχώρου. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να βρω τα όρια του υπολογιστικού νέφους, του cloud computing. Και πολύ θα ήθελα να πιστέψω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι θα δημιουργήσουμε 2,5 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης το 2020 και ότι θα έχουμε 160 δισεκατομμύρια ευρώ που θα, πάνε, θα προσταθούν στο ΕΠ μας. Πολύ ωραία όλα αυτά, πολύ ωραία θα ήταν, αλλά δεν θα συμβεί αν δεν φροντίσουμε να έχουμε και τις σωστές ρυθμίσεις ώστε να υπάρχει το ευρωπαϊκό clouding. Μόνο με αυστηρούς κανόνες και νόμους για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ώστε να μην κινδυνεύουν από εγκληματίες. Αν δεν το κάνουμε αυτό λοιπόν, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νέφος. Ο κύριος Μπάντεν το είπε πριν, σκεφτόσαστε τα email σας. Να, έχω την ενημέρωση εδώ στο iPhone μου και στο iPad μου. Ε, σκεφτείτε τι γίνεται με τις φωτογραφίες σας, εγώ σκέφτομαι τι γίνεται και με τις τραπεζικές μου συναλλαγές. Γιατί όλες ε, οι τράπεζες ε, συνεργάζονται με τον ΕΦΟ σήμερα. Ασφαλιστικές εταιρείες που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τη διευθύνσή σας, να προσθέσετε πληροφορίες στο προφίλ σας, στην ασφάλεια αυτή online. Όλα αυτά γίνονται online. Ε, πού πάνε αυτά τα δεδομένα, πού τα αποθηκεύουν. Η κυρία Χετβέλτα αναφέρθηκε πριν και στο θέμα της υγείας. Εγώ δεν θα ήθελα να μπορεί οποιοδήποτε να κοιτάξει τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την υγεία μου και σίγουρα όχι μια τρίτη χώρα. Το cloud computing είναι μια δραστηριότητα βασισμένη στις Ηνωμένε Πολιτείε ή αλλού, σίγουρα όχι στην Ευρώπη. Και δεν θα είναι αν δεν αφήσουμε τις δικές μας επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν το νέφος. Με την υπόθεση PNR και με τη συμφωνία TFTT, ξέρουμε ότι μεταβάζονται δεδομένα μας στις Ηνωμένε Πολιτείες. Άλλοι το θεωρούν καλό, άλλοι κακό. Το γνωρίζουμε ότι συμβαίνει. Με το cloud computing όμως δεν το γνωρίζουμε. Και δεν το αντιλαμβανόμαστε επίσης. Τώρα για να προστατευτούν οι πολίτες από τους εγκληματίες, από κυβερνήσεις, τα κράτη κτλ. Τρία πράγματα πρέπει να φροντίσουμε. Είναι το hardware, το software, αλλά υπάρχει και ένα τρίτο. Είναι η νομοθεσία. Και εδώ είναι που είναι ο δικός μας ο ρόλος. Γιατί αν δεν υπάρχει η κατάλληλη νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ώστε να είναι υποχρεωμένες και οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις μέσα στην Ευρώπη να φροντίσουν το cloud να γίνεται μέσα στην ευρωπαϊκή δικαιοδοσία και πιθανά άλλο. Θα ήθελα στο Στρασβούργο κατά πάσα πιθανότητα ε, το Μάρτιο να έχουμε μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Και αν έχετε σκεφτεί λίγο τα πράγματα αυτά, αν έχετε νέες ιδέες, πείτε τις μου και θα ετοιμάσω ένα σχέδιο, σχέδιο, σχέδιο, ένα δηλαδή προ-προ σχέδιο ουσιαστικά, να σας παρουσιάσω τον Μάρτιο για να μπορέσουμε πάνω σε αυτό να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σαν. Ευχαριστώ. Ε, ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Κάποιες παρατήρησεις. Ναι. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Well, I want to thank... Uh, Θέλω να ευχαριστήσω τη Γιούντιθ για την προσέγγιση της. Δεν έχω καμιά δυσκολία με την προσέγγιση αυτή. Νομίζω ότι το υπολογιστικό νέφος, που για μένα είναι ιδιαίτερα νεφελώδες, και που φαίνεται ότι μπορεί να έχει πολλά πλέον εκτήματα για τις επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και κίνδυνος από τη χρήση του υπολογιστικού νέφους. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον έλεγχο και την λογοδοσία για την δικαιοδοσία μεταφοράς δεδομένων. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Από τη δική μας πλευρά λοιπόν, από την πλευρά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, θα πρέπει να βασιστούμε στην αρχή ότι οι τεχνολογικές πρόοδοι δεν θα πρέπει να διαβρώνουν τα δικαιώματα των πολιτών και να γίνονται όλα αυτά σε, βάθ, σε βάρος της ε, ιδιωτικότητας των πολιτών. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί και να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία και να υπάρχουν σαφείς κανόνες για λόγοδοσία και να διατηρηθούν τα δικαιώματα της προστασίας των καταναλωτών. Εγώ προσβλέπω στη δυνατότητα να εργαστούμε μαζί με τη Γιούντιτ για αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε κύριε Τριανταφυλλίδη. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο θέλουν να λάβουν το λόγο. Έχοντας ακούσει την ε, παρουσίαση της γνωμοδότησης της εισηγήτριας. Κομισιόν, ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο επικεφαλής μονάδας στην DigiConnect για το υπολογιστικό νέφος. Και θα ήθελα να προσφερθώ στην εισηγήτρια και στα μέλη της Επιτροπής. Μπορούμε να σας δώσουμε οτιδήποτε υποστήριξη θέλετε για την προετοιμασία της γνωμοδότησής σας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η ΛΥΜΠΕ έχει δώσει μεγάλη έμφαση και μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το σημαντικό θέμα και νομίζω ότι και οι συνάδελφοί μας στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη θα είναι έτοιμοι και αυτοί να σας υποστηρίξουν. Έχω συναδέλφους πίσω μου από το τμήμα της DG ε, Δικαιοσύνης που αφορά τις συμβάσεις. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω ότι μία από τις προκλήσεις του υπολογιστικού νέφους είναι ότι αντί τα δεδομένα να είναι υπό τον έλεγχό μας περνάνε σε ένα χώρο που δεν έχει κανείς άμεσο έλεγχο, τίθενται σε ένα υπολογιστή που βρίσκεται στην άλλη άκρη του διαδικτύου. Ένα από τα κέρια θέματα βέβαια είναι η έλλειψη ελέγχου, πώς θα το διαχειριστούμε το θέμα αυτό αφενός. Από την άλλη πλευρά υπάρχει τεράστιο δυναμικό και σημαντικά πλέον εκτήματα που μπορεί να, αντιμετωπι... να αποκομίσει κανείς. Ξέρω ότι η Λίμπε ενδιαφέρει κυρίως για τους κινδύνους αλλά όταν εξετάσετε το θέμα αυτό θα πρέπει να εξισορροπήσετε αυτούς τους κινδύνους έναντι των ευκαιριών που δίδει το υπολογιστικό νέφος. Και εδώ πάλι πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες, να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για να μπορέσει κανείς να εκμεταλλευτεί τα θετικά στοιχεία χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη πολλές τεχνικές τις οποίες υποστηρίζουμε με τα ερευνητικά μας προγράμματα στην DigiConnect που σας επιτρέπουν να αντιμετωπίσετε κάποια από τα προβλήματα που αναφερθήκαν στην απογευματινή συζήτηση. Μπορεί κανείς να σπάει σε κομμάτια τα δεδομένα, ώστε κανείς δεν μπορεί να βάλει, κοντά, να βάλει μαζί όλα αυτά τα διάφορα στοιχεία. Και υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν να διατηρηθεί η κρυπτογράφηση των δεδομένων. Υπάρχουν τεχνικές για να αντιμετωπιστεί ο τρόπος με τον οποίο κρυπτογραφούν τα στοιχεία όταν διαβιβάζονται και όταν ε, <clears throat> αποθηκεύονται, ώστε να μπορεί να γίνει ασφαλής επεξεργασία τους. Υπάρχουν πολλά πράγματα και τα κάνουμε όλα αυτά για να αναπτύξουμε νέες τεχνικές για τα θέματα αυτά. Οι ανησυχίες τώρα για την πρόσβαση των διοκτικών αρχών είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό στην ανακοίνωση της Επιτροπής και ο κύριος Μπάουντεν αναφέρεται σε αυτό. Νομίζω ότι δεν ήταν απόλυτα ακριβή τα στοιχεία που έδωσε. Αναφέρθηκε σε non-papers για συζητήσεις που είχαν να κάνουν με την συνολική συμφωνία αμοιβαία αρρωγή, αλλά δεν έχει υπερατωθεί ακόμα αυτή η διαδικασία. Είναι ένα από του κύριου δρόμου που ακολουθεί η Κομισιόνα για να εξασφαλίσει την κατάλληλη προστασία σε ό,τι αφορά διεθνεί μεταφορέ δεδομένων και την πρόσβαση των διοκτικών αρχών. Είμαι λοιπόν διαθέσιμος για μια συζήτηση με την εισηγήτρια για το πώς ακριβώς λειτουργούν όλες αυτές οι διατάξεις, γιατί νομίζω ότι οι σημερινές παρά παρατη... παρουσιάσεις δεν έλαβαν υπόψη ορισμένε λεπτομέρειε που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα προβλήματα. Δεν θα πω περισσότερε λεπτομέρειε, απλώ ήθελα να πω ότι πολλά από τα θέματα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε στον τομέα αυτό θα αντιμετωπιστούν με συμβατικέ ρήτρε που είναι πολύ σημαντικέ για μα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανεί να προστατευτεί ως ε, πάροχος υπηρεσιών και χρήστης υπηρεσιών στον υπολογιστικό νέφος και ως καταναλωτής. Και ένας από τους χώρους στους οποίους η DigiConnect και η DigiJustice θα εργαστεί είναι να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε καλύτερα τι είδους συμβόλαιο παίρνει κανείς όταν είναι καταναλωτής κάποιος μιας υπηρεσίας στο υπολογιστικό νέφος και να εξασφαλίσουμε ότι είναι λογική δίκαια και διάφανη. Δεν ξέρω λοιπόν αν οι συνάδελφοί μας από την ε, Γενική Διεθνής Δικαιοσύνη θέλουν να πούνε κάτι για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά, γιατί η γνωμοδότηση της ομάδας του άρθρου 29 υπογραμμίζει αυτό το θέμα και υπάρχει αυτή η <clears throat> υποστήριξη που μπορεί να δοθεί σε εσά μέσω των συμβατικών ρητρών που θα συγγραφούν όταν κανείς ξεκινάει μια υπηρεσία. Τα περισσότερα λοιπόν στοιχεία αναφέρονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σε περισσότερα λεπτομέρεια με την εισηγήτρια ή με οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπής σας που ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Η Ιρλανδική Προεδρία θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Εάν όχι. Βλέπω ότι ο κύριος Μπάουντεν θέλει να σχολιάσει. Αν είσαστε σύντομος μονάχα και θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Παρακαλώ. Και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε να κάνω μια σύντομη απάντηση σε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρία στοιχεία μονάχα θέλω να αναφέρω. Η τεχνική του sharding, του θρηματισμού, έχει να κάνει μονάχα με την αποθήκευση, αλλά δεν είναι προστασία για την παράλληλη επεξεργασία στο υπολογιστικό νέφος. Δεύτερον, η δυνατότητα να επεξεργάζεται κανείς ε, κρυπτογραφημένα στοιχεία οι τεχνικές αυτές είναι μία ένα δισεκατομμύριο φορές πιο αργές από την κανονική επεξεργασία. Δεν υπάρχει βιώσιμη τεχνική για τα θέματα αυτά και σε σχέση με το non-paper για τι διαπραγματεύσεις Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωση. δεν έχω πιο πρόσφατα δημόσια έγγραφα, αν υπάρχουν κάποια δημόσια έγγραφα και είναι ενθαρρυντικά, θα ήθελα πράγματι και εγώ να ξέρω. Ευχαριστώ. Κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά, βεβαίως και εγώ θέλω να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ για την προσφορά σας. Αλλά θέλω να κάνω μία ακόμα παρατήρηση για την κρυπτογράφηση. Αντιλαμβάνομαι ότι πέρα από τις παρατηρήσεις του κ. Biden, καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει για την κυβερνοεγκληματικότητα. Αλλά η κρυπτογράφηση δεν θα μας προστατεύσει ε, στην, ε, από τρίτες χώρες οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μας. Δηλαδή μπορεί να είναι μια λύση, αλλά δεν είναι λύση για ολόκληρο το ζήτημα αυτό. Τώρα για την προστασία δεδομένων και τις σχετικές συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε ακόμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όντως δεν μπορούμε να κρίνουμε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα και γιατί θα πάρει πολύ χρόνο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προτιμούσε τι συμφωνίε για το PNR, για το TFTT και τα λοιπά, για την άκτα ίσως. Όλα αυτά θα ήθελε πάρα πολύ να έχουν ε, τελειώσει πριν καταλήξει σε μια γενικότερη συμφωνία για τα ε, δικαιώματα όσον αφορά τον ιδιωτικό βίο και την προστασία των δομένων των πολιτών. Υπάρχει δηλαδή πολιτικός λόγος από πίσω γιατί δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία με τις ΗΠΑ για την προστασία δεδομένων. Και έρχομαι σε αυτό που έλεγα και στην αρχή, μια κατάσταση win-win από την οποία όλοι να έχουν να κερδίσουν. Αν δεν οριοθετήσουμε καλά την υπόθεση αυτή, πάντα θα είναι πιο φτηνά βέβαια είτε η επιχείρηση είτε η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί το υπολογιστικό νέφος για να πουλήσει είτε στις ΗΠΑ είτε σε άλλες χώρες αλλά για να υπάρχει ασφάλεια υπάρχουν πολλά βήματα να γίνουν. Μπορεί να μην αποτελεί αντικείμενο τη συζήτησή μας εδώ στη Λίμπε, αλλά πιστεύω ότι δεν, ε, μάλλον ότι θα βοηθήσουμε την οικονομία μας μόνο εφόσον έχουμε το δικό μας ευρωπαϊκό νέφος με την κατάλληλη νομοθεσία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ συζήτηση είχαμε για το cloud computing. Φαίνεται όντως νεφελώδης ο καιρός. Αναμοδαρμένα ύψη. Και θύελα. Εν πάση περιπτώσει, θα επανέλθουμε. Σύντομα μένουν ακόμα διαδικαστικά ζητήματα έτσι, που πρέπει να λυθούν μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών, διαμάχε δηλαδή για το ποιο είναι πιο αρμόδιο για αυτό το θέμα. Όταν θα έχουν επιληθεί αυτά τα διαδικαστικά, τότε θα έχουμε και προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ όλου σα για τι παρουσιάσει σα, για τι ερωτήσει σα, του προσκεκλημένους μα. Πολύ ενδιαφέρουσα και η συζήτηση που είχαμε. Τώρα δεν βλέπω τον εισηγητή για το επόμενο θέμα. Σε πέντε λεφτά. Α, να νάτι. Η κυρία Μάκιντάιρ. Έρχεται. Πάνω στην ώρα. Τι έγινε, ήρθατε με αλεξίπτωτο εδώ. Πάνω στην ώρα φτάσατε. Προσγειωθήκατε. Μισή ώρα τώρα. Θα είναι και το τελευταίο θέμα για σήμερα το απόγευμα. Αύριο θα συνεχίσουμε στις 9, έτσι. Πρόκειται για την προστασία του νομίσματος, του ευρώχαρτου νομισμάτων και κερμάτων από την παραχάραξη. Δεν πρόκειται μόνο για το ενιαίο νόμισμα της νομισματικής ένωσης, αλλά πρόκειται και για ένα διεθνές νόμισμα. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες που γίνονται από κλιματικές οργανώσεις να παραχαράσουν το ευρώ. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει καταπολέμηση τέτοιων ε, προσπαθειών. Υπάρχει πρόταση της 5ης Φεβρουαρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οδηγία όσον αφορά την προστασία του ευρώ. Στα πλαίσια του ποινικού δικαίου για να προστατεύσουμε το ευρώ. Να μην έχουμε πλαστά νομίσματα. Δηλαδή η κυρία Μάκεντάιρ είναι η συγκεντριά μας και θα μας τα πει όλα αυτά, αλλά προηγουμένως η κυρία Νάτσεν από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης θα μας παρουσιάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είσαστε εδώ? Ναι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Mike, the mic, Mrs. Nutson. Yes, please. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται πολύ που μας δίνεται την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε αυτό το θέμα. Είναι πρότασή μας της 5ης Φεβρουαρίου. Κυρία Ρέντινγκ, ο Επίτροπος ε, Σέμετα επίσης το παρουσίασαν. Η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ έτσι κι αλλιώς, θα το παρουσιάσει στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης αρχές Μαρτίου. Όπως ε, είπαμε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην αυθεντικότητα των χαρτονομισμάτων και των νομισμάτων, οι επιχειρήσεις, οι πολίτες επίσης. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη λοιπόν στο ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι όσοι βρίσκονται με ένα πλαστό νόμισμα, όσο και αν καλό προαίρεται είναι, ποτέ δεν θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Δηλαδή θα μπορέσουν να το ανταλλάξουν με ένα γνήσιο όπως είπε και ο πρόεδρος, εδώ τίθεται θέμα οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται στην παραχάραξη. Είναι εύκολη από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει μια διαδικασία αρκετά περίπλοκη που χρησιμοποιεί το οργανωμένο έγκλημα. Φυσικά κάθε χαρτονόμισμα ευρώ και κέρματα έχουν διάφορα σημεία ασφάλειας και γι' αυτό επειδή δηλαδή το ευρώ συγχρόνω είναι και ένα πετυχημένο νόμισμα, γι' αυτό και αποτελεί ε, αντικείμενο επιθέσεων από τους παραχαράκτες. Επειδή χρησιμοποιείται πάρα πολύ στις διεθνείς συναλλαγές. Το 2002 διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ μετά δηλαδή από την εισαγωγή του νομίσματος. Και σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έχουν εντοπιστεί. Πολύ περισσότερο στο 2012 ε, χαρτονομίσματα τα οποία αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία και ακριβώς όπως είπαμε χρησιμοποιείται μια περίπλοκη τεχνολογία από τις εγκληματικέ οργανώσεις ο εντοπισμός τους γίνεται όλο και πιο δύσκολος. Η Ευρωπόλ είπε ότι υπάρχει μια τάση για αύξηση της εγκληματικότητας σε αυτό το επίπεδο. Είναι μια απειλή που θα παραμείνει, που θα αυξηθεί και όλα στα επόμενα χρόνια από ό,τι φαίνεται. Ανακαλύπτονται διάφορα τυπογραφία και, άλλη, και άλλα εργαστήρια όπου γίνεται η παραχάραξη του ευρώ. Χρησιμοποιείται σε 17 χώρες, 340 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον στόχος Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε να καλύψουμε τις ρυθμιστικές μας αδυναμίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα συμφέρον που είναι κοινό για όλους μας. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Είπα λοιπόν για το ευρώ, γιατί έχει μεγάλη σημασία, αλλά πρέπει να σας πω επίσης ότι η νέα μας πρόταση θα εφαρμόζεται, θα έχει να κάνει δηλαδή και με άλλα νομίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο με το ευρώ. Καλύπτει η πρότασή μας το ευρώ, αλλά καλύπτει και άλλα νομίσματα. Κάτι το οποίο πορεί βέβαια από τη σύμβαση της Γενέβας του 2009 που αναφέρεται στη μη διάκριση. Οπότε δεν κάνουμε εμείς διάκριση στο επίπεδο προστασίας ανάμεσα στο ευρώ και τα άλλα νομίσματα που χρησιμοποιούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 83.1 είναι η νομική μας βάση, η οποία μιλάει για την παραχάραξη μέσων πληρωμής. Δεν αναφέρεται δηλαδή σε συγκεκριμένο νόμισμα. Το επίπεδο προστασίας λοιπόν θα εφαρμόζεται και στο ευρώ και στα άλλα νομίσματα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε πρόκειται για χώρες που είναι opt-in ή opt-out. Ήδη όμως υπάρχουν πολλά μέτρα διοικητικά, κατάρτισης κλπ. που ήδη έχουν εισαχθεί και εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφεύγεται η παραχάραξη. Από πλευρά ποινικών ε, μέτρων, σα είπα, υπάρχει η Σύμβαση της Γενέβη που αναφέρει τι κυρώσει και υπάρχει και κάποια προσέγγιση στην, στις νομοθεσίες των χωρών μελών. Υπάρχει μια απόφαση πλαίσιο επίσης του 2000 που εισάγει ορισμούς και προβλέπει κυρώσεις. Αλλά έχει παλιώσει, είναι 13 ετών. Την είχαμε δηλαδή πριν καν να έχουμε το ευρώ. Συνεπώ τα μέτρα που προβλέπονται από την απόφαση αυτή πλαίσιο δεν είναι τα κατάλληλα. Η αποτροπή δεν είναι αρκετά αποτελεσματική και δεν έχουμε πετύχει και τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Δεδομένου ότι έχουμε τη ζημιά των 500 εκατομμυρίων που σας είπα. Επιπλέον, οι αποφάσεις πλαίσιο δεν έχουν την ίδια ισχύ όπως θα έχει μελλοντική οδηγία. Βέβαια εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο ε, επίσης στην κάθε χώρα. Το καλό με την οδηγία είναι ότι έτσι μπορούν να καλυφθούν οι διαφορετικές αδυναμίες στις διάφορες χώρες. Η νέα μας πρόταση πρέπει να σας πω ότι δεν διαφέρει βέβαια ριζικά από την απόφαση πλαίσιο, καλύπτει αδυναμίες φυσικά, και να... αλλά βασίζεται στην παλιά αυτή απόφαση πλαίσιο. Διευκρινίζει κάποια σημεία και προσθέτει λεπτομέρειες. Κρατέ τους ίδιους ορισμούς που θα γνωρίζετε από την απόφαση πλαίσιο. Και βάσει της νομικής μας βάσης 83.1 καθορίζουμε και ελάχιστους κανόνες για κυρώσεις. Η πρόταση συνολικά θα έλεγα ότι έχει ως στόχο τα μέσα εκείνα και τα εργαλεία που έχουν ήδη εντοπιστεί από διάφορες διαβουλεύσεις που είχαμε μέχρι τώρα για να ενισχυθεί η προστασία του ευρώ. Υπήρξε ευρεία διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, κρατημέλη, ομάδες εμπειρογνωμόνων και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φυσικά και όλοι μας βοήθησαν να καταλήξουμε στα μέτρα τα οποία προτείνουμε εδώ. Το στοιχείο κλειδί πάντως είναι η έννοια της πιο ε, των πιο αποτελεσματικών εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές υπεύθυνε για την επιβολή του νόμου. Δεύτερον, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ε, τα νομίσματα τα οποία ε, κατάσχονται, τα παραχαγμένα δηλαδή, φροντίζουμε τι θα γίνουν μετά ώστε να μην κυκλοφορήσουν φυσικά πάλι, είναι σημεία τα οποία καλύπτονται πιο πολύ από την Γενική Διεύθυνση Όλαφ. Και το τρίτο νέο στοιχείο είναι οι κυρώσεις, που εμείς θέλουμε να είναι πιο αποτελεσματικές, έτσι ώστε να είναι τα μέτρα αυτά πιο αποτρεπτικά ανώτατες ποινές τόσο για την ε, παραγωγή όσο και για τη διανομή νομισμάτων κύβδηλων και να υπάρχουν ελάχιστες κυρώσεις κάθε φορά. Όσον αφορά τις κυρώσεις, καλό θα ήταν εδώ πέρα να πούμε ότι αυτό περιλαμβάνεται ήδη στην απόφαση πλαίσιο. Μιλάμε για 8 χρόνια. Το επαναλαμβάνουμε και στη νέα πρόταση και αντικατοπτρίζει και την κατάσταση που ισχύει στα κράτη-μέλη που θεωρεί την παραχάραξη πολύ σοβαρό αδίκημα και τιμωρείται αυστηρά. Θέλουμε να επεκτείνουμε το επίπεδο αυτό και στη διανομή τώρα. που δεν καλύπτονταν ε, μέχρι τώρα από κυρώσεις μετά από έγκλημα που είχε αυτό τον νότο των 8 ετών αλλά και η διανομή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να γίνει μέσα ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από διάφορα κανάλια. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να καταπολεμήσουμε και τη διανομή. Γιατί οι δράστες φυσικά και θέλουν να κυκλοφορούν ε, τα νομίσματα αυτά εύκολα. Οπότε προσθέτουμε και την διανομή κύβδηλων νομισμάτων και συμπεριλαμβάνεται πια και αυτή στις κυρώσεις μας. Και για τις ε, τρίτες χώρες αναφερόμαστε, είναι ένας τρόπος αυτός να εντοπίζουμε τις διόδους μέσω των οποίων τα κύβδηλα αυτά νομίσματα μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον ε, έχουν παραχθεί εκτός. Πιστεύουμε ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το όλο ζήτημα των ε, σχετικών ε, δραστηριοτήτων. Βάζουμε και μία ελάχιστη κύρωση φυλάκισης έξι μηνών και για την παραγωγή και για την διανομή των πλαστών ε, νομισμάτων με διάφορες ρήτρες ασφαλείας. Για μας είναι και αυτό αποτροπή και ο λόγος είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο αυστηρό επίπεδο για να μπορούμε να εμποδίζουμε έτσι αυτού του είδους το παράπτωμα. Οι ανώτατες ποινές, βλέπετε, διαπιστώσαμε ότι δεν φτάνουν. με τις ελάχιστες πιστεύουμε ότι κάνουμε την αποτροπή ακόμα πιο ισχυρή. Είναι πιο αποτρεπτικό να ξέρεις ότι θα καταλήξεις στη φυλακή από το να έχεις πρόστιμο. Πάντως, βάζουμε και διάφορες δίτες ασφαλείας και λέμε ότι προβλέπονται αυτές οι ελάχιστες ποινές για τις πιο σοβαρές, τα πιο σοβαρά δικήματα, παραγωγή και διανομή και μόνο στις σοβαρές ε, περιπτώσεις, δηλαδή όταν εμπλέκεται ε, σημαντικός όγκος χρημάτων. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις ελάχιστες ποινές που προβλέπουν, που είναι από το 0 μέχρι τα 10 χρόνια. Οι διαφορές αυτές καταλαβαίνετε ότι μπορεί να οδηγήσουν το κάθε δράστη να πηγαίνει εκεί όπου ξέρει ότι δεν προβλέπονται ποινές ή ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές. Θέλουμε λοιπόν το μέτρο αυτό να είναι αποτρεπτικό και σημαντικό, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι κυρώσεις είναι και ανάλογες του αδικήματος. Δημιουργούμε λοιπόν ένα σύστημα διαφοροποίησης της ποινές και έχουμε διαφορετικά κατόφλια εισάγουμε την ε, έννοια του μικρού αδικήματος κάτω από 5 πτέσματος, κάτω από 5.000 για παράδειγμα, προβλέπουμε πρόστιμο. Λαμβάνουμε υπόψη μας ε, δηλαδή το μέγεθος του παραπτώματος. Υπάρχει διαβάθμιση λοιπόν. Μετά μιλάμε για ποσά 5 με 10.000 ευρώ όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβλέψουν σε αυτή την περίπτωση κάποιο είδους φυλάκιση ε, που ίσως θα μπορούσε να είναι και κάτω από 6 μήνες με πρόστιμο. Και βέβαια προβλέπουμε και την άλλη κατηγορία για πάνω από 10.000 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις που όταν είμαστε πάνω από 10.000 οι χώρες θα πρέπει να προβλέψουν οπωσδήποτε μία ελάχιστη ποινή. Πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η αρχή της εθνικής νομοθεσίας, δηλαδή ότι οι εθνικοί νόμοι ισχύουν για την εκτέλεση και για την επιβολή της ποινής. Αλλά κάθε φορά θα υπάρχει ένα ελάχιστο και ένα ανώτατο. Αν υπάρχουν ελαφρυντικά, τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν και χαμηλότερη ποινή του εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν είναι η πρώτη φορά που ε, πιάνε το δράστης ή αν πρόκειται για ανήλικο. Αυτό είναι στη διακριτική ευχαίρεια της χώρας μέλους. Μπορούν δηλαδή να επιλέξουν εναλλακτικέ ποινές ή να ελευθερώσουν τον δράστη νωρίτερα κτλ. κτλ. Μπορείτε να καταλήξετε στα συμπεράσματά σας, λέει ο Πρόεδρος, διακόπτοντας την ομιλήτρια. Γιατί μιλάτε 20 λεπτά, οπότε σταματήστε παρακαλώ. Γιατί έχουμε και την εισηγήτρια, έτσι. Έχετε δίκιο και συγγνώμη γιατί μιλάω πολύ. Τα μέτρα αυτά παρέχουν ισορροπημένη πρόταση που θα συμπληρωθεί με μια σειρά μέτρων ανακριτικού χαρακτήρα και μέτρα διήμευσης που θα σχολιάσει συνάδελφος από την Όλαφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Η Όλαφ. Η κυρία Χόφμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τη συνάδελφο για την εισαγωγή. Να σας πω ποια είμαι. Είμαι διευθύντρια πολιτική στην Όλαφα, στο τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη σημαντική αυτή η πρόταση. Όπως ξέρετε και η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη και η Όλαφ είναι η... στην εμπροστοφυλακή της πρότασης αυτής. Όπως είπε η κυρία Κνούτσεν, θα σταθώ σε δύο συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την παραχάραξη. Ένα, την διάσταξη για τα ουσιαστικά ανακριτικά εργαλεία άρθρο 9 και δεύτερον την ε, μεταφορά ε, των ε, κατασκευέντων χρημάτων. Νέα στοιχεία σε σχέση με την απόφαση πλαίσιο του 2001. Τα δύο αυτά θέματα συμπεριλήφθηκαν ρητά στην πρόταση μετά από αίτημα των εμπλεκόμενων στο εθνικό επίπεδο της Τράπεζας και της Europol για να μειωθεί, μειωθούν τα κενά που είχαν διαπιστωθεί. Τούτο έγινε μετά από μακρά διαβούλευση με ερωτηματολόγια, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων κτλ. Τεράστια διαβούλευση δηλαδή. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην πράξη και που αναφέρονται στη, και αναφέρθηκαν στη διαβούλευση σχετίζονται με την διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών και περιγράφω την κατάσταση εντάχει. Σε κάποια κράτη-μέλη, στην Ιταλία για παράδειγμα, δεν υπάρχουν ανακριτικά εργαλεία διαθέσιμα που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για οργανωμένο έγκλημα και ειδικά στοχοθετημένα για την αντιμετώπιση της παραχάραξης, δηλαδή ε, μυστικοί πράκτορες, μυ, μυστικοί ε, αστυνομικοί κλπ. Επίσης, όταν ξεκινά η έρευνα σε ένα κράτος μέλος όπου βρίσκονται τα χαρτονομίσματα, δεν μπορεί να συνεχιστεί σε άλλη χώρα όπου δεν υπάρχει εκεί όπου εμφανίστηκαν τα, τα χαρτονομίσματα, εκεί που κυκλοφόρησαν δηλαδή τα χαρτονομίσματα, γιατί δεν υπάρχουν στο δεύτερο κράτος τα ανακριτικά μέσα που απαιτούνται. Η λύση προβλέπεται στο άρθρο 9. Ζητείται από όλα τα κράτη-μέλη να έχουν τα ίδια ουσιαστικά ε, ανακριτικά μέσα στη διάθεσή τους για να καταπολεμήσουν την παραχάραξη. Αυτό δεν είναι καινούριο για σας. Θα δείτε αντίστοιχα, αντίστοιχες διατάξεις ε, στην οδηγία για την πρόληψη της διακίνησης ε, της εμπορίας ανθρώπων του Απριλίου του 2011. Το δεύτερο σημείο τώρα. Το δεύτερο παραθυράκι που εντόπισαν οι εμπλεκόμενοι ήταν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υποχρέωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο δυνατότητα με τον κανονισμό 1338 του 2001 να μεταβιβάζονται τα κατασχεθέντα ευρώ, παραχαραγμένα ευρώ, κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών για τεχνική ανάλυση για να μπορούν να εξετάσουν και να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άλλα παραχαραγμένα χατονομίσματα στην κυκλοφορία. Υπάρχουν περιπτώσεις μάλιστα όπου οι δικαστικές αρχές δεν αρνήθηκαν να δώσουν αντίτυπα ε, να δώσουν δείγματα αυτού του, αυτών των παραχαραχθέντων νομισμάτων πριν ολοκληρωθεί η δίκη. Αυτό είναι σημαντικό κατά απόψή μας. Η μεταφορά των, των παραχαραγμένων μετά το τέλος της δίκης έχει πολύ μικρή αξία. Συχνά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις δίκες, παίρνουν χρόνο πριν φτάσει ας πούμε πριν ε, προσαρμοστούν οι αρχές στα νέα εργαλεία, στις νέες ε, πρέσες. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Η λύση ποια είναι, να προβλέπουμε υποχρέωση, όχι δυνατότητα, η, να μεταβιβάζουν οι δικαστικές αρχές ή να δίνουν πρόσβαση τουλάχιστον στα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης των Τραπεζογραμματείων, το CNAX, Coin National Analysis Centers for Coins, CNAC τα λέμε εμείς, δείγματα των ε, κατασχεθέντων ε, νομισμάτων και χαρτονομισμάτων για ανάλυση. Στο άρθρο 10 της πρότασης. Αυτά ήταν τα δύο σημεία που θέλω να σχολιάσω. Συνοψίζοντας, η επιστροφή προτείνει ότι αυτό είναι σημαντικό βήμα μπρος για να υποστηρίξουμε την ε, καταπολέμηση της πλαστογράφησης του, της παραχάραξης του ευρώ και των άλλων νομισμάτων. Τα στατιστικά δεν σα τα δώσω, αλλά πιστεύουμε ότι η πρόταση έρχεται στη σωστή στιγμή. Είναι φτιαγμένη ακριβώς όπως ε, χρειάζεται για να εξυγχρονίσουμε το υφιστάμενο πλαίσιο, την απόφαση πλαίσιο δηλαδή, και παρέχει νέα στοιχεία στηριζόμενη στο κεκτημένο και η Κομισιόν και η Όλαφ ε, στηριζόμαστε στην υποστήριξή σας, στην υποστήριξη και της κυρίας η εισηγήτριας και του Κοινοβουλίου ολόκληρου για να έχουμε ένα στιβαρό εργαλείο για την προστασία του ενιαίου νομίσματος αλλά και των άλλων νομισμάτων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τις δυο σας. Και τώρα προδίνω το λόγο στην κυρία Μάκεντάιρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Κομισιόν και την Όλαφ για τις παρουσιάσεις τους. Όλοι τα χαιρετίζαμε μέτρα τα οποία αντιμετωπίσουν την παραχάραξη χαρτονομισμάτων που φυσικά έχουν αρνητικό αποτέλεσμα για όλες τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από το αν το Βασίλειο έχει το δικό του νόμισμα η παραχάραξη των ευρώ αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσθέσω επίσης θα ήθελα τα μέτρα για την προστασία αναφέρονται σαν μέτρα προστασίας του ευρώ και άλλων νομισμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πράγματι πρόσφορο να επικαιροποιήσουμε την απόφαση πλαίσιο Όπω είπε η Κομισιόν, το ευρώ δεν υπήρχε όταν θεσπίστηκαν οι πρώτοι κανονισμοί. Και... και είμαι έτοιμη να συνεργαστώ με τους κοιότητες εισηγητές για να έχουμε μια χρήσιμη έκθεση. Απλώς θα ήθελα να με ένα σημείο όπου η Κομισιόν ενδεχομένως θα μπορούσε να επανέλθει. Πιστεύω προσωπικά ότι η ανείχνευση είναι το πιο σημαντικό αποτρεπτικό στοιχείο αυτός που τουλάχιστον ισχύει στη δική μου χώρα. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτό που λέει η Κομισιό ότι έχουμε μια μέγιστη, ε, ένα μέγιστο πρόστιμο, μια μέγιστη ποινή, αλλά δεν έχουμε ελάχιστη ποινή και γι' αυτό το λόγο, επειδή η μέγιστη ποινή δεν απέδωσε αποτέλεσμα, έχουμε τώρα μια ελάχιστη ποινή. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια στοιχεία τους οδηγούν στο να θεσπίσουν μια κατώτατη ποινή. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Ένας άλλος τομέας. Και αυτό πάλι ένα μικρό σημείο, το άρθρο 8, 8.1β. Εδώ αναρωτιέμαι για την πρακτική εφαρμογή. Λέει ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη δικαιοδοσία του για τους ε, αδικοπράκτες όταν είναι πολίτες τους, υπηκοοί τους. Μα οι αστυνομίε δρούν σε ένα κράτος και φυσικά έχουν δικαιοδοσία για τα δικήματα που λαμβάνουν χώρα στη δική τους χώρα. Έχουμε και το ευρωπαϊκό ένταλμα το οποίο επιτρέπει να δικαστούν άτομα ακόμα και αν δεν βρίσκονται στο μέρος όπου διέπραξαν το αδίκημα αυτό. Αλλά αυτό είναι σαν να λέμε ότι κάθε χώρα πρέπει να είναι υπεύθυνη για αδικήματα που έκαναν οι πολίτες της και σε άλλες χώρες. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί συμπεριλαμβάνεται αυτή η ρήτρα. <clears throat> Ίσως θα μπορείτε να με βοηθήσετε να καταλάβω πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Γενικά όμως εγώ χαιρετίζω το γεγονός ότι επικαιροποιούμε αυτές τις ρυθμίσεις και τις φέρνουμε στον νέο αιώνα και έχω πλήρη υποστήριξη και προσβλέπω στο να συνεργαστώ και με τους συναδέλφους για να έχουμε μια εποφελή έκθεση. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. <clears throat> Βλέπω ότι και η κυρία Ματιό θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Το ΕΛΚ είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την πρόταση οδηγίας όσον αφορά την παραχάραξη και την πλαστογραφία των ε, ευρώ και των άλλων νομισμάτων πρόκειται συχνά για μια διασυνοριακή εγκληματική δραστηριότητα. Η παραχάραξη φυσικά πλήττει τον πολίτη, γιατί είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Φτάνει κανείς να πληρώσει το κρέας του στο κρεοπολείο και δίνει ένα χαρτονόμισμα και του λένε «Όχι, είναι πλαστό» φυσικά ο πολίτης χάνει γιατί δεν του δίνει κανένας ε, ένα γνήσιο χαρτονόμισμα σε αντάλλαγμα αυτού. Όπως επίσης είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό στοιχίζει 500 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Είναι καλή πρόταση λοιπόν να αρμονίζει την προστασία του ευρώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκαθιστά επίσης την Σύμβαση της Γενέβης και την αρχή της μη διάκρισης εφόσον προστατεύονται από την ίδια οδηγία και τα άλλα νομίσματα που κυκλοφορούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολύ καλή αλληλεγγύη πράγματι και βάζει έξι μήνες και επιτρέπει οι δράστες να διώκονται βάσει του ευρωπαϊκού ε, Σύμφωνη Europol, Eurojust. Είναι αλήθεια ότι δεν το είχαμε αυτό ακόμα και είναι πολύ καλό που το έχουμε τώρα. Έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν η Επιτροπή λέει ότι απογοητεύτηκε από τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα για την παραχάραξη, γιατί γενικά για τα πλαστά προϊόντα ή ειδικά για την παραχάραξη. Όντω υπήρχαν διατάξει στα κράτη-μέλη για την παραχάραξη που προφανώ δεν ήταν ε, ότι καλύτερο. Αλλά γενικά για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας, των πλαστών μάλλον προϊόντων, εδώ υπάρχουν ε, προδιαγραφές που είναι πιο κατάλληλες. Αλλά γενικά με τα πλαστά προϊόντα βλέπουμε ότι δεν προχωράμε αρκετά. Οπότε γι' αυτό θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενικά σας απογοητεύουν τα αποτελέσματα από την καταπολέμηση των πλαστών προϊόντων. Ωραία. Ακούστηκαν ερωτήσεις, πολύ συγκεκριμένες. Πριν τελειώσουμε, λίγα λεπτά για να μας απαντήσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε χαιρόμαστε πολύ που ακούμε ότι η πρόταση αυτή έτυχε καλής αποδοχής στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και προσβλέπουμε επίσης και στη συνεργασία με την κυρία εισηγήτρια και τις σκιώδους εισηγητές. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την καλή υποδοχή της οποίας έτυχε η πρότασή μας. Ήθελα απλώς να πω προς την κυρία Μακιντάε που φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε και περαιτέρω. Να πω για το ερώτημά της για την ε, δικαιοδοσία. Νομίζω ότι μίλησε για το άρθρο 8 παράγραφος 1. Β. Κυρία Μακιντάε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό το θέμα υπήρξε και στην ε, απόφαση πλαίσιο και εγγράφεται και στη σύμβαση της Γενέλης. Επομένως ε, ενσωματώνουμε τη Σύμβαση της Γενέβης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αν θέλετε μπορούμε να τα συζητήσουμε πιο λεπτομεριακά αγότερα. μικρόφωνο, Θα συνεχίσουμε στις 9 αύριο.